Chers collègues, je vous propose de prendre place en m'excusant de ces 10 minutes de retard. Ζητώ συγγνώμη για τα 10 λεπτά καθυστέρησης. Λοιπόν, α περάσουμε στη συνεθέτηση τη ημερήσια διάταξη. Να σα πω ότι υπάρχουν τρει αλλαγέ. Καταρχήν το σημείο 19 που αφορά την ψηφοφορία για τη συμφωνία με το Συμβούλιο για την Ελεύθερη Κυκλοφορία των Εργαζομένων, την έκθεση της κυρίας Μπάουερ, θα αναβληθεί και θα συζητηθεί μετά το σημείο 22, δηλαδή μετά από την ψηφοφορία για το σχέδιο γνωμοδότησης της κυρίας Γιασλοβιέσκα για τους ε, εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας. Ε, το, η έκθεση της κυρίας Μάκιντάρ για τη δημιουργία κατάλληλου ε, περιβάλλοντος ώστε οι επιχειρήσεις να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης θα αναβληθεί για την έκτακτη μα συνεδρίαση που θα γίνει στις 3 Φεβρουαρίου το, στο Στρασβούργο. Τέλος, το σημείο 23 για την ανταλλαγή απόψεων για τα διδάγματα που πρέπει να αντιληφθούν στο πλαίσιο των ε, διαπραγματεύσεων για το PDP θα οδηγήσει σε σύνταξη γνωμοδότησης, διότι εντωμεταξύ η Επιτροπή Προπολογισμών έχει πάρει έγκριση για να συντάξει έκθεση πρωτοβουλίας και άρα λοιπόν ε, έχουμε χρόνο να ετοιμάσουμε σχέδιο χρονοδότηση σε έφετο χρόνο για αυτή την έκθεση πρωτοβουλία. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει, λοιπόν, ε, θα σε εγκρίνουμε, εγκρίνεται μάλλον η μερίσια διάταξη όπω τοποποιήθηκε. Σα ευχαριστώ και περνάμε στο σημείο 2 ανακοινώσει τη Προέδρου. Όσον αφορά την συνεδρίαση τη Επιτροπή Απασχόληση 12 και 13 Φεβρουαρίου, σα λέω ότι αυτή η συνεδρία θα ξεκινήσει στις 3 ε, στις 12 Φεβρουαρίου και κατά συνέπεια το πρωινό της 12 Φεβρουαρίου ακυρώνεται. Τώρα, για την διερμηνία που δεν χρησιμοποιείται, θα πρέπει να σας πω ότι στη συνεδρία της ομάδας εργασίας de la commission ECON της Επιτροπής ΕΚΟΝ για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Η Ισπανική διερμηνία δεν χρησιμοποιήθηκε γιατί ο κύριος Γκουτιέρης Πιώτο δεν συμμετείχε στη συνεδρίαση χωρίς να ενημερώσει προηγουμένως τη γραμματεία και άρα αυτό δεν μας επέτρεψε να ακυρώσουμε την εν λόγω διερμηνία. Επιπλέον, η γαλλική διερμηνία δεν είχε ζητηθεί, διότι ο κύριος Γκουτιέρης Πριώτο είχε συγκεκριμένα ζητήσει την ισπανική διερμηνία ως εισηγητής της Επιτροπής Απασχόλησης, πράγμα το οποίο περιόριζε τις δυνατότητες διερμηνίας. Ε, τρίτο σημείο, ως ήθιστε, ε, για την ηλεκτρονική ε, αναμετάδοση των εργασιών μας στο ίντερνετ. Μπορείτε όλα αυτά να τα δείτε μέσω της εφαρμογής e-meeting και μέσω ίντερνετ. Σημείο 3. Προτείνω την έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων της 14ης και 18ης Νοεμβρίου. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις μέχρι το τέλος της συνεδρίασης θα θεωρήσουμε ότι εγκρίνονται τα πρακτικά αυτά. Και φτάνουμε έτσι στο σημείο 4 της ημερήσιάς μας διάταξης. Πρόκειται για την εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης για την έκθεση που συντάσσει η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού για το θέμα των εργαλείων που έχουν ε, ε, χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση ε, της αποτελεσματικότητας των δαπανών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για τους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας. Μετά από την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου 25 κάθετος 2012. Και γι' αυτό το σημείο δίνω το λόγο στην εισηγήτριά μας, Ντανούτα Γιασλοβιέσκα, η οποία θα μας ενημερώσει για τις ε, τροπολογίες που κατετέθησαν επτά από την ίδια και με βάση τις οποίες συμβιβαστικές, ε, μάλλον υποβλήθηκαν και επτά συμβαστικές τροπολογίες. Κυρία Ισηγήτρια, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Δεδομένου ότι είχαμε μείωση του αριθμού του παραγωγικού δυναμικού πέρυσι, θα πρέπει να ξεπίσουμε περισσότερο τους μεγαλύτερες ηλικιές εργαζόμενους ε, στο Ευρωπαϊκό Ταμείο είχαμε για την περίοδο 75 ε, ευρώ 2007, για την περίοδο 2007-2013. Επιπλέον, τα κράτη-μέλη είχαν 117 λειτουργικά προγράμματα. 60 από αυτά είχαν ή άμεσα ή έμεσα ως ε, αποδέκτες τους μεγαλύτερης ηλικίας εργαζομένους. Ε, με βάση την έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου το 2012, ούτε τα κράτη-μέλη, ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι σε θέση να ε, ενημερώσουν για το πώς οι μεγαλύτερες ηλικίες εργαζόμενοι ε, χρησιμοποίησαν ή υποφελήθηκαν από τα κονδύλια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Ούτε μπορούμε να πούμε πόσες ενέργειες του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και πόσες επεμβάσεις ήταν αποτελεσματικές ε, και βελτίωσαν τους μεγαλύτερους εργαζόμενους να εμπλουτίσουν τις δεξιότητες τους ή να βρουν καλύτερη θέση απασχόλησης. Τώρα προτείνονται κάποιοι μηχανισμοί για τη βελτίωση της παρακολούθησης ε, και του ελέγχου των κονδυλίων ε, που είναι αφιερωμένα για τους, είναι αφιερωμένα Έχουμε 1 τροπολογίες. Από αυτές ε, συντάξαμε 7 συμβαστικές τροπολογίες, προσπαθώντας να καλύψουμε τις περισσότερες από τις τροπολογίες των συναδέλφων. Η συμβεστική τροπολογία α, ε, στα στοιχεία που δυσκολεύουν τους ηλικιωμένους να βρουν δουλειά, αναφέραμε τις, μικρό, τις λιγότερες απασχόλησης και την ε, αύξηση της ανταγωνιστικότητας μεταξύ των εργαζομένων. Επίσης, η απόφαση για παραμονή στην αγορά εργασία μετά το συντάξιμο όριο ηλικία εναπόκειται στον εργαζόμενο. Συμβαστική τροπολογία Β. Πρώτα απ' όλα στην συμβαστική τροπολογία Β επισημάναμε τη διαφορά στη... μεταξύ ανδρών και γυναικών σε ό,τι αφορά του ηλικιωμένου εργαζομένους. Γιατί 54% ε, είναι το ποσοστό ε, για τους άνδρες, ενώ για τις γυναίκες είναι πολύ μεγαλύτερο. Δηλαδή, πιο μεγάλες ηλικίε ε, γυναίκες που παραμένουν στα αγορά εργασίας είναι πολύ λιγότερες από τους άντρες. Επίσης, ως αιτία αυτής της α, ε, μικρής παραμονής στην αγορά εργασίας των ηλικιωμένων είναι λίγες δεξιότητες ή δυσκολίε στη συμφιλίωση οικογενειακή και επαγγελματική ζωή. Στη συμβαστική τροπολογία Γ επισημάναμε το γεγονό ότι τα κονδύλια του ΕΚΤ για το 2007-2013 ήταν 8% του προπολογισμού και στην κατάσταση, στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να ελέγχεται πολύ καλύτερη αποτελεσματικότητα των κονδυλίων. Συμβαστική τροπολογία Δέλτα, πρώτη παράγραφος, λέμε ότι οι πληροφορίες για τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, καθώς και οι πληροφορίες για τις δαπάνες ε, που έχουν τέτοιο σκόπο, θα πρέπει να είναι προσιτές ε, ε, δημοσίως, να δημοσιεύονται στο διαδίκτυο και επίσης να συνοδεύονται με στοιχεία για τις διαφορές μεταξύ των φύλων. Στο ε, θέλουμε, εκτός από τις πληροφορίες για το πώς οι εργαζόμενοι βελτίωσαν τις δεξιότητές τους χάρη στα κονδύλια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και αύξησαν τις ικανότητές τους, θέλουμε ε, και πληροφορίες για το πώς ηλικιωμένοι έλαβαν μέρος σε τέτοια προγράμματα, πόσοι από αυτούς απέκτησαν νέες δεξιότητες και πόσοι βρήκαν μία θέση εργασίας. Και επίσης θέλουμε να συγκεντρώνονται στοιχεία και για τα δύο φύλλα. Στην έκτη συμβαστική πρόταση, στην πέμπτη παράγραφο, λέμε ότι θα πρέπει να είναι αποτελεσματικά τα προγράμματα του ΕΚΤ και να είναι προσανατολισμένα στα αποτελέσματα για να μπορούμε στο μέλλον να λάβουμε τεκμηρωμένες αποφάσεις. Η τελευταία συμβαστική τροπολογία αφορά την 7η παράγραφο και μιλά για την ανάγκη συνεχούς παρακολούθησης πολιτικής για τους ηλικιωμένους στα πλαίσια της διαβίου κατάρτισης και της ενεργούς γύρανσης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις και ηγετρίες για τη συνεργασία τους και ευελπιστώ ότι στην ψηφοφορία θα υπερψηφιστούν όλες οι συμβαστικές τροπολογίες. Σας ευχαριστώ. Merci, euh, Phil Et puis, qui a qui Αυτά. κύριος Μπένιον. Θα είμαι πολύ σύντομος, γιατί νομίζω πως η συγκίτρια εργάστηκε πάρα πολύ αποτελεσματικά και εμείς στην ομάδα ALDE υποστηρίζουμε όλες τις προτινόμενες συμβιβαστικές και τις περισσότερες τροπολογίες ε, που είναι εκτός των συμβιβαστικών. Δεν υποστηρίζουμε την τροπολογία 25, αλλά Μπορούμε να στηρίξουμε την 31 αν η προφορική η τροπολογία της εισηγήτρες είναι αποδεκτή και αυτά μόνο έχουμε να πούμε για την ώρα. Ευχαριστώ. Ελιζαμπέτ Μωράν Σαρτιέ, πολύ σύντομα Κυρία Πρόεδρε, για να ευχαριστήσω την εισηγήτριά μα για την εργασία τη, διότι όλα τα σημεία τα οποία έθιξε τονίστηκαν και στην εργασία μα για την περίοδο 2014 με 2020 και είναι σημεία που θέλουμε να βελτιώσουμε στο μέλλον. Ευχαριστώ λοιπόν που ήρθατε και στηρίζετε την εργασία μας για το πολιετές. Merci. est a Ce n'est pas le cas. Je donne la parole à notre pour conclure. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ θερμά τους και όλους ε, για τη συνεργασία τους. Στον κύριο Φιλ Μπένιον θα ήθελα να πω ότι για την τροπολογία 31 για τις αναλύσεις ε, στην αγορά εργασίας. Οι αναλύσεις αυτές ε, γίνονται σε εθνικό επίπεδο γιατί δεν έχουμε ομοιόμορφο σύστημα. Και έτσι ε, τουλάχιστον θα έχουμε πληροφορίες ανακράτος μέλος. Ελπίζω στο μέλλον να έχουμε πολύ πιο ενοποιημένες στατιστικές και μεθόδους. Γι' αυτό θα ήθελα να θερμαπαρακαλέσω τους φιλελεύθερους να δεχτούν τελικά την τροπολογία μου 31. Bien. Euh, sur cette Ωραία. Από αυτές τις βάσεις θα ψηφίσουμε στις 23 Ιανουαρίου, ε, δηλαδή αύριο. Πράγμα που θα επιτρέψει στην Επιτροπή Προπολογισμού να λάβει υπόψη την ε, νομοδότησή μας αυτή στην ψηφοφορία της περνάμε στο σημείο 5. Εξέταση των συμβαστικών τροπολογιών που δεν ξέρω πόσες είναι. Ο κύριος Γκουτιέρης Πιουριέτο δεν είναι εδώ, πράγμα που δεν είναι πρώτη φορά. Η κυρία Μάκιντάιρ είναι εδώ, είναι εδώ. Να μην μου λέει μετά κανείς που εξετάσαμε την έκθεση της κυρίας Μακιντάρ, τη απουσία των σκιωδών ε, εισηγητών. Οι συντονιστές μου επιτρέπουν λοιπόν να εξετάσουμε την έκθεση της κυρίας Μάκιντάρ, ενώ δεν είναι εδώ κανένας από τους σκιώδεις, εκτός από τον κύριο Τεμπάκερ. Ναι, ωραία λοιπόν. Να πάμε στο σημείο 6. Αλλά ζητώ από τους ε, πολιτικούς υπαλλήλους να μεριμνούν ώστε όταν οι, τα μέλη πρέπει να είναι παρόντες, να είναι παρόντες, ώστε να μην αποδιοργανώνεται η εργασία των υπόλοιπων ευρωβουλευτών και των ε, υπόλοιπων υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένων και των διερμηνέων. Λοιπόν, εξετάζουμε τις 42 συμβιβαστικές τροπολογίες για την έκθεση της κυρίας Μάκινταερα. Πριν να της δώσουμε το λόγο, θα ήθελα να υποδείξω κάποιες δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε σε αυτή την έκθεση και που έχουν να κάνουν, που έχει τίτλο πώς μπορεί να συμβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη διαμόρφωση ευνοϊκού περιβάλλοντος για τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις και νεοσύστατες επιχειρήσεις. Πρόκειται για μια έκθεση πρωτοβουλίας που συζητήθηκε και αποφασίστηκε με τη συμφωνία των συντονιστών μετά από τρεις φορές όπου εξετάστηκε το αντικείμενο της έκθεσης, για το λόγο ότι από τη μια πλευρά η Επιτροπή ΙΜΚΟ μόλις είχε συντάξει έκθεση πρωτοβουλίας για ένα παρόμοιο θέμα και επειδή ε, χρειάστηκε να παρεύουμε τρεις φορές ε, στους συντονιστές για να φτάσουμε σε έναν τίτλο για την έκθεση πρωτοβουλίας που θα επιτρέψει να στοχεύσουμε στις συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων στον τομέα. Ωστόσο, η αρχική έκθεση της εισηγητρίας συμπεριλάμβανε σύμφωνα με την εμπειρογνωμοσύνη της γραμματείας της Επιτροπής μας και όχι σύμφωνα με τη δική μου γνώμη, πολλές παραγράφους που δεν ήταν αρμοδιότητα της Επιτροπής μας. Και όπως το πράττουμε συχνά, επιστήσαμε την προσοχή της ε, συντάκτριας στο γεγονός ότι αυτές οι, παράγραφοι θα έπρεπε να τροποποιηθούν για να είναι αποδεκτές και όχι να θεωρήσουμε ότι αυτές δεν μπορούσαν να γίνουν αποδεκτές εξ αρχής. Την ίδια δυσκολία αντιμετωπίσαμε πολλές τροπολογίες που υποβλήθηκαν από τους συναδέλφους συμπεριλαμβανομένων τροπολογιών που στόχο είχαν να καταργήσουν ένα τμήμα των αρχικών παραγράφων της εισηγήτριας και που αν καταργούσαμε αυτές τις παραγράφους θα καταργείτο και η αρμοδιότητα της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Ορισμένοι, όπως ο κ. Κρούτσμαν, με κατηγόρησαν ότι διοργάνωσα εγώ αυθαίρετα και μερικώς την αποδοχή αυτών των παραγράφων. Δεν δέχομαι αυτήν την επίκριση για ιστορικούς λόγους που σας θύμισα και διευκρινίζοντας ακόμη μια φορά ότι δεν ήμουν εγώ που ε, κρίνα, αλλά ακολούθησα τη γνωμοδότηση που μου δόθηκε από τη γραμματεία μας και από όσο γνωρίζω η γραμματεία αυτής της Επιτροπής δεν μπορεί ε, καθόλου να κατηγορηθεί για ότι δεν είναι μερόληπτη από πολιτικής άποψης. Δεν σε επιτρέπεται εξάλλου να προβαίνει σε πολιτικές αξιολογήσεις ή εκτιμήσεις. Ελπίζω λοιπόν ότι θα μπορέσουμε τώρα να μιλήσουμε με χρήσιμο και επικοδομητικό τρόπο για την έκθεση της κυρίας Μακιντάρ, γιατί στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τις συμβαστικέ ε, παραμένουν πολλά προβλήματα και γι' αυτό το λόγο στην έναρξη των εργασιών μας ήδη σας υπέδειξα ότι δεν θα μπορέσουμε να ψηφίσουμε αύριο για αυτή την έκθεση. Αυτά έχω, κάθε, έχω πλήρη εμπιστοσύνη στην εισηγήτριά μας ώστε να επικρατήσει ε, να επικρατήσουν και να επανέλθουν στην καρδιά αυτής της έκθεσης οι αρμοδιότητες της Επιτροπής μας και έτσι ώστε η συζήτηση να είναι χρήσιμη και σκόπιμη με σεβασμό στις αρμοδιότητες μας διότι δεν θέλω να κάνουμε σε άλλες επιτροπές αυτό που δεν μου αρέσει να μας χάνουν. Κυρία Εισηγήτρια, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και να αρχίσω με ευχαριστίες πρώτα προς τους συναδέλφους μου που συνεργάστηκαν ε, για το φάκελο αυτό και χαίρομαι που αναβλήθηκε για την 3η Φεβρουαρίου η ψηφοφορία γιατί θα μας επιτρέψει ο χρόνος αυτός να εξετάσουμε κάποια κρεμή θέματα. Είχαμε 276 τροπολογίες, τόσες υποβλήθηκαν για την έκθεσή μου. Καταλήξαμε δε σε 40 περίπου συμβιβαστικές τροπολογίες που συνέπτυξαν 157 συνολικά διάφορες τροπολογίες. Γι' αυτό είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη και ευχαριστώ τους συναδέλφους μου διότι μπορέσαμε μέσα στις συμβαστικές τροπολογίες να συμπτύξουμε τόσα πολλά πράγματα. Νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε επί των συμβαστικών, αν και μείνει ακόμα δουλειά να γίνει. Ορισμένοι συνάδελφοί μου έχουν ζητήσει και άλλες αλλαγές θα κάνω κάθε δυνατή προσπάθεια για να περιλάβω τα σχόλιά τους και θα διανύμω κάποιες νέες προτάσεις θα εξετάσω και οτιδήποτε οποιοδήποτε επιχείρημα που λέει ότι εκφεύγουμε των αρμοδιοτήτων, των αρμοδιοτήτων μας και θα κοιτάξω ώστε να γίνουν σεβαστοί οι κανόνες περί αρμοδιοτήτων. Τώρα, σε δύο συμβαστικές τροπολογίες, την ΔΕΛΤΑ, ΔΕΛΤΑ, DD, την οποία θα διαγράψουμε, διότι δεν μπορέσαμε να συμφωνήσουμε. Τελικά θα ψηφίσουμε τις επιμέρους τροπολογίες και η άλλη είναι η Z, όπου πάλι δεν φαίνεται να μπορούμε να συμφωνήσουμε και θα επανέλθουμε στις αρχικές τροπολογίες. Πέραν όμως αυτών των δύο, νομίζω ότι δεν έχουμε άλλα σημαντικά εμπόδια. Θα έλθω λοιπόν σε επαφή με τους συναδέλφους μου μεμονωμένα για να ζητήσω την υποστήριξή τους και μιας και έχουμε περισσότερο χρόνο, ελπίζω να μπορέσω την επόμενη Τετάρτη απόγευμα να οργανώσω την τελική πια συνάντηση των συντονιστών με την ελπίδα ότι όλοι θα μπορέσουν να συμφωνήσουν με τις ε, τελευταίες και τελικές αυτές ε, συμβαστικές προτάσεις. Η Ήτρε έχει ένα κανόνα 50 για την έκθεση αυτή και υπάρχουν ορισμένες παράγραφοι από ε, τη δική τους γνωμοδότηση που περιλαμβάνονται στην έκθεση. Υπάρχουν όμως και ορισμένες παραγραφοί που δεν είναι ούτε ε, αρμοδιότητα της Ήτρε ούτε άλλης επιτροπής παρά μόνο έκον. και επειδή η ΕΚΟΝ δεν έκανε τίποτα, δεν νομίζω ότι τα θέματα αυτά, τα αντικείμενα δηλαδή των ε, παραγράφων αυτό της ΕΚΟΝ, θα πρέπει να μπουν στο δικό μας κείμενο. Και ελπίζω οι συντονιστές να με ενισχύσουν. Αναμένω τα σχόλια των συναδέλφων και θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι όλες τις συντονίστες και συντονιστές για την συμβολή τους και ελπίζω να μπορέσουμε να συνεργαστούμε στο ε, θετικό αυτό πνεύμα συνεργασίας το οποίο κατήσχησε μέχρι τώρα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρία Ισηγήτρια. Συμφωνώ με την αξιολόγησή σας για τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ήτρε. για την οποία ούτε και τα ίδια τα μέλη της Επιτροπής αυτής δηλαδή δεν σεβάστηκαν απόλυτα τα όρια αρμοδιοτήτων τους. Αν και προηγουμένως έκανα λάθος αυτή είχε κάνει προηγουμένως την εργασία αυτή σε προηγούμενη έκθεση πρωτοβουλίας με παρόμοιο θέμα και όχι, όπως λάθος είπα πριν, η Οικονομική Επιτροπή. Τώρα, το λόγο θα δώσω στον Φίλιπ Ντεμπάκερ. Ευχαριστώ, καθώς επίσης ευχαριστώ και την εισηγήτρια για τη σκληρή δουλειά που έχει κάνει έως τώρα λάβαμε τις πολλές προτάσεις συμβαστικών τροπολογιών και όπως είπα έκανε καλή δουλειά. Είδαμε ότι και πολλές από τις δικές μας τροπολογίες περιλήφθηκαν τελικά. Τώρα, για τη συμβαστική ε υπάρχει τώρα ένα μέρος το οποίο προστίθεται στο αρχικό κείμενο για βιώσιμες δημόσιες επενδύσεις. Είναι σημαντικό εδώ να υπάρξει μια σύνδεση και με τις δημόσιες προμήθειες. Γιατί αυτό είναι ένα εργαλείο και απέναντι στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να μπορούν να συμμετέχουν δηλαδή στις δημόσιες προμήθειες γιατί με τον τρόπο αυτό θα υπάρξει και ανάπτυξη και κάποια δημιουργία απασχόλησης αν ληφθεί υπόψη αυτό. Για τη συμβαστική Q με το αρχικό κείμενο που περιλαμβάνει και φορολογικά κίνητρα. Δεν ξέρω αν ε, έγκυται αυτό στις αρμοδιότητες επιτροπής μας για την συμβαστική π. θέλουμε να αφαιρεθούν οι λέξεις or information set distributed γιατί προκαλούν κάποια σύγχυση. Φαίνεται να υπάρχει επιλογή μεταξύ του one-stop shop από τη μια μεριά και μεταξύ των περιφερειακών κέντρων πληροφοριών από την άλλη μεριά. Πρέπει όμως να ευθυγραμμιστούμε τις διατυπώσεις του Enterprise Europe Network για την συμβαστική μη μη ε, να είμαστε κάπως πιο ουδέτεροι σε ό,τι αφορά τα φύλλα γιατί ε, οι όροι που χρησιμοποιούνται εκεί αφορούν και τα δύο φύλλα. Δηλαδή το προσδόκιμο ε, ζωής κλπ. Έλαβα κι εγώ ένα ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σχετικά με το μη παραδεκτό ορισμένων τροπολογίων. Είναι περίεργο να ζητείτε να διαγράψει ένα τμήμα του κειμένου επειδή είναι μη παραδεκτό. Εν πάση περιπτώσει έχουμε ακόμα μερικές τροπολογίε, Θα συζητήσουμε και με τη Γενική Γραμματεία για να δούμε αν μπορούμε να διατηρήσουμε ορισμένε από τι τροπολογίε που αρχικά κρίθηκαν μη παραδεκτές. Θα δούμε αν μπορέσει να προκύψει κάποια λύση. πάντω, οι συνάδελφοί μου και εγώ αναμένουμε την συνέχιση της μέχρι τώρα θετικής συνεργασίας. Σας ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον Σέρζιο Αγκουτιέρες Πριέτο. Ευχαριστώντας τον ε, που βρήκε τελικά το δρόμο προς την αίθουσα. Αν και λυπούμε που δεν ήταν στην ώρα του για να συζητήσουμε ως δεύτερο σημείο το δικό του. Τώρα, σε σχέση με αυτά που είπε ο Φιλίπ Τεμπάκερ. Αν κάνουμε πράγματα που δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητές μας, είναι λογικό να κρίνονται ως μια παραδεκτά Αν η αρχική έκθεση σε μία παράγραφο λέει, τώρα παράδειγμα λέω, ότι οι επιχειρήσεις, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις πρέπει να είναι πιο ανταγωνιστικές. Μα αυτό δεν είναι δική μας αρμοδιότητα. Δεν είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόλησης. Οπότε από τη στιγμή που δεν εμπίπτει ένα θέμα στις αρμοδιότητες μας, η, η συγγήτρια τροποποιεί την αρχική παράγραφο και λέει η επιχειρήσεις πρέπει να γίνουν πιο ανταγωνιστικές για να δημιουργήσουν τις απασχόλησης, τότε μπίπτει στις αρμοδιότητές μας και άρα γίνεται παραδεκτή. Τώρα, αν θέλετε να διαγραφεί αυτό και να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης, επανερχόμαστε στην αρχική κατάσταση, δεν ε, καλύπτει δικές μας αρμοδιότητες και άρα ξαναγίνεται μη παραδεκτή τροπολογία. Νομίζω ότι είναι πολύ ορθός αυτός ο τρόπος και ε, ευθύς ε, για να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα, ουδέτερος και αμεροληπτικός. Ε, δεν ικανοποιούμε ούτε την αριστερά ούτε την δεξιά. Αλλά αν σταματήσουμε εκεί την παράγραφο δεν είναι πια παραδεκτή η τροπολογία. Και ο λόγος τώρα στον Σέρζιο Γκουτιέρες Πρέτο. Καταρχήν να ζητήσω συγγνώμη από τα μέλη της Επιτροπής και το Προεδρείο. Από τη στιγμή που κάποιος αισθανθεί μια διαθεσία θα πρέπει να είμαστε κάπως ελαστικοί για να το τροποποιούμε την ημερήσια διάταξη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Μακεντάιρ για τις συμβαστικές τροπολογίες που κατέθεσε. Γιατί στην αρχική της έκθεση ήταν ε, πολύ μακριά από την ε, προσέγγιση των σοσιαλιστών και θα ήταν σχεδόν αδύνατο να την εγκρίνουμε, αλλά στο μεταξύ σημειώσαμε πρόοδο. Και στην πρώτη ανταλλαγή απόψεων και με τις τροπολογίες η κατάσταση εξελίχθηκε και ευχαριστώ την εισηγήτρια που προσπάθησε με τις τροπολογίες να λάβει υπόψη και τις δικές μας ευαισθησίες. Αρχίζει και οριμάζει η κατάσταση, οπότε είμαστε πια σε θέση να υπερψηφίσουμε τις ε, συμβαστικές τροπολογίες. Θα πρέπει όμως να διευκρινίσουμε μερικές από αυτές, γιατί εξακολουθούν να απάδουν από την ε, θέση των σοσιαλιστών. Για παράδειγμα, στη συμβαστική τροπολογία D το έμεσο εργασιακό κόστος, που είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στις επιχειρήσεις, επιμένουμε η μνή αυτή να αντικατασταθεί από κάτι πιο σφαιρικό και κάτι που βρίσκεται πιο κοντά στην πραγματικότητα, τις τρέχουσες πάνες, για παράδειγμα. Γιατί το έμεσο εργασιακό κόστος είναι αντίστοιχο με το ενεργειακό κόστος για τις επιχειρήσεις. Νομίζω ότι η δική μας πρόταση είναι καλύτερη γιατί διευρύνει την έννοια αυτή. Επίσης έχω καταθέσει την τροπολογία 171 για να προσθεθεί στο τέλος της έκθεσης. Προβλήματα θα έχουμε και με τη συμβαστική τροπολογία α, από ό,τι βλέπω. Αλλά αν αντικατασταθεί το τελευταίο τμήμα της συμβαστικής τροπολογίας ε, Α. Ε, από την τροπολογία 220 της κυρίας Κορνέλησεν θα βελτιωθεί η συμβαστική λύση και έτσι θα μπορέσουμε να την υπερψηφίσουμε. Πρόβλημα έχω με την συμβαστική τροπολογία ΣΕΣΕ που μιλάει για τον αντίκτυπο που έχουν κάποιες διατάξεις ε, ε, υγείας ε, και προστασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις. Πάντως είμαστε στη διάθεση της και πρόθυμοι για συνεργασία προκειμένου να διευκρινίσουμε κάποια σημεία της έκθεσης. Γιατί δεν νομίζω ότι η νομοθεσία για την υγεία και την προστασία των εργαζομένων είναι αρνητική ή δημιουργεί προβλήματα στην απασχόληση. Πρόβλημα έχουμε και με την τροπολογία FF που μιλάει για την απόσπαση των εργαζομένων, posting. Οπότε θα καταθέσουμε μία μικρή πρόταση αναδιατύπωσης για να μπορέσουμε να την υπερψηφίσουμε. Αυτά και ευχαριστώ την εισηγήτρια, αναγνωρίζω τις προσπάθειές της γιατί δείχνουν την προθυμία της ε, για συνεργασία και αναζήτηση συμβαστικής λύσης. Ευχαριστώ πολύ. Άλλος κανείς δεν έχει ζητήσει τον λόγο εκ των συναδέλφων μας. Ίσως όμως η Κομισιόν επιθυμεί να λάβει τον λόγο. Ναι, όχι, δεν έχω το όνομά σας, αλλά αν θέλετε ευχαρίστως. Εμείς είμαστε ικανοποιημένες από αυτή την έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας γιατί θα επιτρέψει στις ε, επιχειρήσεις να δημιουργήσουν απασχόληση και είναι σημαντικό για την ε, βιομηχανική πολιτική. Η Κομισιόν σήμερα ενέκρινε νέο ανακοινοθέν για την βιομηχανική πολιτική με κύριο μήνυμα ότι η Ευρώπη χρειάζεται επιγόντως να βάλει τις βάσεις για την ανάπτυξη μετά την κρίση, μια αναζωογόνηση της οικονομίας. Και στη βάση αυτή, και καθώς και των σχεδιασμών του 2010 και 2012, θα βασίσουμε τις περιοτεραιότητες της βιομηχανικής πολιτικής για να αποδώσουν αποτέλεσμα. Äh, Ο Προεδρεύων, ευχαριστώ. Η συγγήτρια θα πάλι τον λόγο. Μέχρι τώρα άκουσα μόνο καλά λόγια. Έχετε βεβαίως ακόμη λίγη δουλειά να κάνετε, νομίζω όμως ότι το αποτέλεσμα θα είναι θετικό. Έχετε το λόγο κυρία μου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι πράγματι ευγνώμων για την υποστήριξη που έλαβα από τους ε, άλλους εισηγητές. Είναι και μια σημαντική εμπειρία για μένα η σύνταξη αυτή τη έκθεση. Τώρα για τον κύριο Ντεμπάκερ. Σας υποστηρίζω απολύτως σε αυτό που λέτε για τη σημασία των δημοσίων προμηθειών και βεβαίως θα θέσω το θέμα. Τα φορολογικά κίνητρα νομίζω θα είναι δύσκολο να περιληφθούν διότι πάμε έτσι και μπαίνουμε στα οικόπεδα της Επιτροπής ΕΚΟΝ. Δεν νομίζω να μπορώ να βοηθήσω πολύ εκεί. Για το Enterprise Europe Network, ναι. Και βεβαίως για τον όρο που αναφέρατε που πρέπει να είναι ουδέτερος όσον αφορά το φύλλο, βεβαίως δεν είναι μόνο για τις γυναίκες. Όρο όρος life balance δηλαδή δεν αφορά μόνο γυναίκες αλλά και τα δύο φύλλα. Σωστό. Σεις κύριε Πρίατο τώρα, βγάλαμε από την συμβαστική TAF τη λέξη labor. Οπότε μιλεί μόνο για έμεσα κόστη. Ελπίζω λοιπόν ότι σας ικανοποιεί αυτό ώστε να μπορέσετε να συμφωνήσετε. Ασφαλώς και θα εξετάσω ξανά την συμβαστική α και επίσης την CC και FF. Και βεβαίως Επαναλαμβάνω ότι χαίρομαι που θα γίνει ψηφοφορία αργότερα, δηλαδή στις 3 Δευτέρου, γιατί αν μπορέσουμε να συναντηθούμε ξανά την επόμενη εβδομάδα, νομίζω ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε κάτι το οποίο θα υποστηριχθεί ευρέω. Χάρηκα επίση που άκουσα θετικά λόγια και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ελπίζω ότι λοιπόν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορέσει να δεχθεί την έκθεσή μου όταν θα την λάβει. Ευχαριστώ. Ο Τόμας Μαν, Προεδρεύων. Νομίζω ότι όντως αξίζουν τον κόπο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ε, εγκύψουμε στα συμφέροντά τους. Άρα δεν θα ψηφίσουμε τελικώς αύριο, το λέω αυτό για όσους ενδεχομένως ήρθαν με κάποια καθυστέρηση, αλλά στις 3 Φεβρουαρίου, 3 Δευτέρου. Σύμφωνα τώρα με την ημερησία διάταξη, θέμα υπαριθμών 6 που μόλις συζητήσαμε τώρα, έρχεται το επόμενο 7. Ο κύριος Γκουτιέρες Πριέτο θα παρουσιάσει την εκθεσή του και θα μπορέσουμε να την συζητήσουμε. Και η επομένη συνάδελφο θα χρειαστεί να περιμένει λίγο ακόμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα, εν συντομία, να ευχαριστήσω πρώτα τους σκιώδης ηγητές για την ε, διαλλακτικότητά τους και το συνεργάσιμο πνεύμα τους. Δεν ήταν εύκολο να καταλήξουμε σε συμφωνία για την έκθεση αυτή. Αφενός είχαμε το πιεστικό χρονοδιάγραμμα. Οπότε θα πρέπει να παρακολουθήσουμε τις προθεσμίες του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και να ψηφίσουμε στην Ολομέλεια του Φεβρουαρίου. Κάτι που μας συρρήκνωσε την προθεσμία για την υποβολή και τη συζήτηση των τροπολογιών. Ευχαριστώ λοιπόν για την συνεργασία τους τους συναδέλφους, γιατί ξεκινούσαμε από διαφορετικά σημεία αφετηρίας και διαφορετικές απόψεις, αλλά είχαμε διπλό στόχο. Θέλαμε ένα στεναρό μήνυμα της Επιτροπής Απασχόλησης και χρήσιμο για την προάσπιση των θέσεων της Επιτροπής μας και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απέναντι στο Συμβούλιο για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και με συμπληρωματικό τρόπο και όχι αντιφατικό σε σχέση με την αντίστοιχη έκθεση της ΕΚΟΝ. Νομίζω ότι πλησιάζουμε όλο και περισσότερο σε μία συμφωνία. Θα πρέπει, όπως είπα και στο παρελθόν, θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι η προσπάθεια να είναι συμπληρωματική δική μας έκθεση σε σχέση με την έκθεση Depacker της Επιτροπής ΕΚΟΝ δεν σημαίνει θα είναι μια έκθεση που απλώς θα μιμείται την έκθεση της ΕΚΟΝ γιατί η κατάσταση στις κοινωνικές υποθέσεις είναι πολύ πιο οξία και χαλεπή σε σχέση με την οικονομική κατάσταση. Επεξεργάστηκα γύρω στις 33 τροπολογίες, συμβαστικές τροπολογίες και βρισκόμαστε στην τελική φάση οριστικοποίησης της διατύπωσής τους, ώστε να καταφέρουμε να ψηφίσουμε αύριο. Πάντως υπάρχει γενική συμφωνία για την έκθεση. Τα περισσότερα προβλήματα τα είχαμε με το παράρτημα. Και επειδή το έχουμε συζητήσει επανειλημμένο στην Επιτροπή, θα ήθελα να είμαι κατηγορηματικός. Ξεκινούσαμε από μια κρατούσα άποψη και σχεδόν συνένεση για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, ότι θέλουμε να κρατήσουμε στην έκθεση τα παραρτήματα αυτό είχαμε αποφασίσει και στην προηγούμενη έκθεση χωρίς κανένα πρόβλημα από καμία πολιτική ομάδα και ξεκινώντας από την ε, θέση του κυρίου Ντεμπάκερ και της ε, έκθεσης ΕΚΟΝ που κατάργησε όλα τα παραρτήματα και τις παραγράφους μας δημιούργησε πρόβλημα. Αυτή η θέση έγινε δεκτή τελικά από τους φιλελεύθερους και φαίνεται ότι και το ΕΛΚ έχει κάποιες αφιβολίες για την αναγκαιότητα μιας τέτοιας πρότασης, δηλαδή της διατήρησης των παραρτημάτων. Εγώ πιστεύω ότι θα ήταν ακατανόητη αυτή η παλινδρόμηση στην προσπάθεια ανάκτησης της δημοκρατικής νομοποίησης η κατάργηση των παραρτημάτων. Και αν τελικά το ΕΛΚ επιδιώξει μία πλειοψηφία για την κατάργηση αυτή των παραρτημάτων. Εμείς θέλουμε να ενισχύσουμε τη δημοκρατική νομοποίηση, όχι να την αποδυναμώσουμε. Και με την κατάρριξη των παραρτημάτων το αντίθετο αποτέλεσμα θα έχουμε, την αποδυνάμωση ουσιαστικά της δημοκρατικής νομοποίησης. Οπότε εγώ ως θα ήθελα να εκφράσω την έκπληξή μου για αυτές τις αφιβολίες που δημιουργήθηκαν και αυτές τις παλιδρομήσεις και θα ήθελα να ζητήσω από τους φιλελεύθερους και το ΕΡΚ να σκεφτούν πολύ προσεκτικά τις συνέπειες ενός τέτοιου μηνύματος ε, προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Ενός μηνύματος ουσιαστικά που θα μας γυρίσει πίσω. Αυτά και ευχαριστώ τους και οδησηγητές για τη συνεργασία. Πιστεύω όμως ότι αν δεν γίνουν ε, κάποιες ε, μεταστροφές στη γνώμη τελευταία στιγμή, θα καταφέρουμε αύριο με μεγάλη πλειοψηφία να υπερψηφίσουμε την έκθεση. Θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Όρη, που το ζήτησε, αλλά θα ήθελα από θεσμική άποψη να επανέλθω στο θέμα αυτό. Η συζήτηση, η ουσιαστική συζήτηση στην δημοκρατία αφορά τους προσανατολισμούς της οικονομικής πολιτικής. Αυτή είναι η κυραχοκοκαλιά των δημόσιων πολιτικών. πέραν κάποιων άλλων δραστηριοτήτων ε, που δεν ανήκουν στις δικές μας αρμοδιότητες. Η συζήτηση αυτή είναι αρκετά ακαθόδης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί μιλούμε για ένα τομέα που εμπίπτει κυρίως σε εθνικές αρμοδιότητες. Το άρθρο 121 της συνθήκης λέει ότι τα θέματα της ε, οικονομικής πολιτικής θα πρέπει να θεωρηθούν από τα κράτη-μέλη ως θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Ενώ το άρθρο 145 λέει κάπως πιο χαλαρά κάτι αντίστοιχο για τις πολιτικές απασχόλησης. Οπότε με αυτή τη βάση οι κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση και οι μείζονες προσανατολισμοί για την οικονομία εντάσσονται στη συνθήκη. Με βάση τις συνθήκες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει για τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση μεγαλύτερες εξουσίες ε, σε σχέση με αυτές που έχει η Οικονομική Επιτροπή για τους μείζονες οικονομικούς προσανατολισμούς. Με την προηγούμενη μου ιδιότητα ως πρόεδρο της Επιτροπής ΕΚΟΝ ε, φρόντισα, με ρίμισα τουλάχιστον, να αναθεωρούνται ιονοί νομοθετικά έγγραφα αυτοί μείζονες οικονομικοί προσανατολισμοί. Και στην αρχή της κοινοβουλευτικής θητείας είχαμε μία αναθεώρηση με τον εισηγητή Τη αντίστοιχη έκθεση τη Επιτροπή Απασχόληση, τον κύριο Ρίρ, και καταφέραμε με τη βοήθεια της Βελικής Προεδρίας να επηρεάσουμε και την διατύπωση των κατευθυντηρίων γραμμών για την απασχόληση. Στα, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και με την ετήσια επισκόπηση για την ανάπτυξη άλλαξαν τα χαρακτηριστικά και το καθεστώς αυτών των δύο θα θυμάστε ότι πριν από λίγο καιρό είχαμε ανταλλαγή απόψεων με τον πρόεδρο της ΕΜΚΟ. Και σήμερα το πρωί φτάσαμε στο τέλος της δεύτερης κοινοβουλευτικής εβδομάδας, που είναι η ευκαιρία για μια διακοινοβουλευτική συζήτηση με θέμα την ετήσια επισκόπηση και την ανάπτυξη. Δυστυχώς το Συμβούλιο δεν ε, έχει δεχτεί όλα τα αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν θα ήθελα όμως να επαναχωρήσουμε σε σχέση με προηγούμενες πρακτικές μας και στη συνέχεια να αρνηθούμε κάτι που βρίσκεται στην καρδιά του κοινωνικού συμβολέου και της διατησίας της οικονομικής πολιτικής. Θα πρέπει τέτοιες εξουσίες μας να τις ε, αξιοποιήσουμε και να τις ασκήσουμε στο έπακρο. Υπάρχουν βέβαια νομικά επιχειρήματα που μιλούν για παραβίαση των συνθήκων ή μία απόλυτη ευθυγράμμιση των συνθήκων. Αν όμως εμέναμε με αυστηρά στο γράμμα της συνθήκης, ελάχιστα θα κάναμε και δεν θα είχαμε καμία συζήτηση για το παραδεκτό των ε, εκθέσεων πρωτοβουλίας, γιατί δεν θα χρειαζόταν καν να κάνουμε εκθέσεις πρωτοβουλίας. Κάθε φορά που εξετάζουμε το θέμα αυτό χρειάζεται να επαναλάβω όλα αυτά τα πράγματα. Πάντως θεωρώ ότι είναι ουσιώδη ζήτημα για τις αρμοδιότητες της Επιτροπής μας, για τις εξουσίες του Κοινοβουλίου και για την διεξαγωγή δημοκρατικής συζήτησης ε, για την οικονομική και κοινωνική πολιτική. Πιστεύω ότι είναι σημαντική η δημοκρατική νομοποίηση για τις πολιτικές αυτές. Ο λόγος τώρα στον Τζαμπαόρη και μετά στη Μαριάν Χάρκιν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ ζητώ το λόγο εξ ονόματος ε, του κυρίου Λόπε Φοντανιέ, που δυστυχώς χρειάστηκε να επιστρέψει στην Ισπανία. Κάναμε πολύ σοβαρές συζητήσεις, προπαρασκευαστικές συζητήσεις για αυτό το θέμα και Εν μέρη, συμμεριζόμαστε την ανάλυση της Προέδρου. Υπάρχουν σίγουρα θετικά στοιχεία στην έκθεση. Και μας καθησυχάζει το γεγονός ότι δίνεται έμφαση στις επενδύσεις στα κίνητρα για την ανάπτυξη, το ρόλο της γυναίκας, τις, τις ποιοτικέ θέσεις απασχόλησης, ε, την ε, συμφιλίωση της ιδιωτικής με την ε, επαγγελματική ζωή, τον ορισμό των τομέων προτεραιότητας και συμφωνούμε και για το γεγονός για την νεανική εγγύηση. Ωστόσο υπάρχουν πολλές δυσκολίες όσον αφορά τις συμβιβαστικέ. Ε, σίγουρα δεν μπορούμε να ε, υποστηρίξουμε την συμβιβαστική ΑΣ, αλλά ούτε και την ε, ΕΝ. Ναι. Και όσον αφορά την B, την Q, την ΡΟ και την S, εμείς είμαστε ακόμα στη συζήτηση. Δεν έχουμε καταλήξει αν θα πούμε ναι ή όχι. Και όσον αφορά τώρα τα παραρτήματα. Θα πρέπει να σας πω ότι εγώ δεν θέτω τόσο πολύ θέματα αρμοδιότητας ή κυριαρχία. Δεν έχουμε ακόμα αποφασίσει. Ας ε, προσπαθήσουμε, προτείνουμε μάλλον να δεχτούμε τη δυνατότητα ε, να υπάρξουν τα παραρτήματα. Είναι κάτι που ήθιστε εφόσον πρόκειται για έκθεση πρωτοβουλία. Ε, δεν είναι κάτι το καινούριο. Αλλά τελικά μετά από ορισμένες συζητήσεις αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε ακόμα να αρνηθούμε κατηγορηματικά. Ήμασταν μάλλον διχασμένοι λοιπόν για αυτό το θέμα και συνεχίζουμε να το συζητάμε. Αυτά έχω να σας πω όσον αφορά τη θέση μας. Thank you, Chair, and... Uh, ευχαριστώ κυρία Χάρκιν. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ τον εισηγητή για την πολύ καλή συνεργασία που είχε μαζί μας κατά τη διάρκεια των ε, διασκέψεών μας. Φτιάσαμε σε συμφωνία σε πολλά θέματα και ήταν πολύ θετική η εργασία. Έχω μόνο κάποια σχόλια όσον αφορά κάποιες συμβιβαστικές. Συμβαστική age, H. Από ό,τι κατάλαβα και θα ήθελα την γνώμη του ησυχητή από αυτού, Καταψηφίστηκε το μήνυμα με επίδομα ανεργία στην Ευρωζώνη, γιατί λέει εδώ πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά από την Κομισιόν να εκπονήσει έγγραφο. Δεν ήταν ο Λόπε αλλά θυμάμαι ότι καταψηφίστηκε στην έκθεση Φερέιρα στην Ολομέλεια. Άρα λοιπόν αυτό είναι πρόβλημα και από ό,τι κατάλαβα και το ΕΛΚΑ έχει το ίδιο πρόβλημα. Στην συμβαστική ΆΗ σας ευχαριστώ και πάλι. Ζητώ να... Ε, είχα ζητήσει μάλλον να ακολουθηθεί η γραμμή της έκθεσης και ε, και αυτό γίνεται σε μεγάλο βαθμό και στηρίζουμε το τελευταίο τμήμα. Να ρωτήσω όμως, γιατί υπάρχει αρκετά μεγάλο κομμάτι νέο κειμένου στην παράγραφο αυτή που ξεκινά ε, με το είναι της άποψης ότι και ολοκληρώνεται υπό την συντονισμό της οικονομικής πολιτικής. Θέλω να ρωτήσω από πού προήλθε, είναι νέο κείμενο, αλλά ίσως να είναι ε, από κάποια παλιότερη έκθεση. Το επόμενο που θέλω να σχολιάσω είναι η συμβιβαστική K. Και πάλι ευχαριστώ τον εισηγητή. Αυτό προέρχεται από το ψήφισμα για την κοινωνική διάσταση και σας ευχαριστώ που το αλλάξατε ώστε να μπορούμε και εμείς να το υποστηρίξουμε. Επίσης για την συμβιβαστική N, ε, θα, μπορεί να κάνουμε κάποια επιπλέον συζήτηση με την ομάδα μας, αλλά βλέπω και πάλι πως ε, αλλάξατε προς την κατεύθυνση που ζητήσαμε ένα κομμάτι του κειμένου και δεν ξέρω πόσο τώρα αυτό θα γίνει δεκτό και συμβαστική ο... Ε, ελπίζω πως θα μπορέσουμε να τη στηρίξουμε γιατί εδώ αφαίρεσατε το νούμερο και έτσι ελπίζω πως θα μπορέσουμε να την υποστηρίξουμε. Θέλω να ρωτήσω για τη συμβαστική Q όπου λέτε και πάλι και αυτό μόνο για να ελέγξουμε ότι είναι σωστό, σωστή διατύπωση. Λέει, σημειώνει πως η ανακοίνωση για το PDP ε, για την της επισκόπηση για την ανάπτυξη του 2014 και τα λοιπά. Δεν ξέρω τώρα αν είναι απόλυτα σωστό. Μήπως θα έπρεπε να είναι οφείλει να είναι ή θα μπορούσε να είναι. Είναι όντως έτσι ή η Κομισιόν λέει ότι θα πρέπει να ειναι ειναι οντω ετσι έτσι. Μπορείτε αυτό να το διευκρινίσετε. Τέλος, και νομίζω ότι οι υπόλοιπε τροπολογίε οι περισσότερε είναι εντάξει. Αν κάπου υπήρχε μια κόκκινη γραμμή, ποια ήταν η L. Α, συγγνώμη γιατί δεν μπορώ να την βρω αυτή τη στιγμή. Εκεί όπου γίνεται λόγος για Θα το βρω σε λίγο. Συγγνώμη. Ευχαριστώ επίσης γιατί στην ε, συμβιβαστική α η ε, χρησιμοποίησατε την έκθεση Μενερόιτεν. DD είπατε, μάλιστα. Έχουμε πρόβλημα στην DD. Το πρώτο κομμάτι είναι εντάξει, λέει καλή την Επιτροπή να αναπτύξει την κοινωνική πτυχή και τα στην ΟΝΕ. Ε, το δεύτερο τμήμα που λέει να επεξεργαστεί περισσότερο το τρόπο εισαγωγή ενό προγράμματος Ευρωπαϊκού Επιδόματος Ενεργείας. Εδώ αυτό ήταν ανέκαθεν κόκκινη γραμμή για μας. Επίσης, στο τέλος ε, της συμβαστικής ή e, το ίδιο θέμα για την αξιολόγηση, το κείμενο θα πρέπει να επανεληφθεί ε, ακριβώς και όσον αφορά τα παρατήματα, ε, κρατούν διαφορετικές απόψεις εντός της ομάδας. Ξέρετε, μας είπαν ότι δεν θα περάσει από την έκονα, αλλά αυτή είναι η δική μας νομοδότηση. Για τη γνώμη μου θα πρέπει να μείνει η δική μας νομοδότηση και έχω δύο παραρτήματα. Στη συμβιβαστική ΙΙ το θέμα είναι αν θα πρέπει να αποσυρθεί η ΕΛ και στην BB αν περιλαμβάνεται η DD που ανέφερα πριν από λίγο που είναι κόκκινη γραμμή για μας, οπότε θα είναι πρόβλημα για μας. Νομίζω πως υπάρχει μεγάλο βαθμό συμφωνίας και δυναμικό για σημαντική συμφωνία αν την ψηφίσουμε αύριο με κάποιες μικροαλλαγές. Ευχαριστώ και πάλι τον εισηγητή για την εξαιρετική του εργασία. Θέλει άλλος κανείς το λόγο? Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, λέει ο κύριος Δεμπέκερ. Και εγώ έχω κάποια σχόλια και να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Ξέρω, εισηγητή τη Επιτροπή ΕΚΟΝ, πόσο δύσκολο είναι να συμβιβάσει κανεί τι διάφορε απόψει. Πολλά δεν βάλουν όταν αποκλίνουν αρκετά μεταξύ του. Το ίδιο και στην ΕΚΟΝ. Έχω και εγώ πρόβλημα. Ελπίζω όμω να έχουμε τελικά δύο επιτροπέ με δύο εκθέσει σαφεί και διαφανεί. Συμφωνώ με τι περισσότερε τροπολογίε. Έχω περίπου τα ίδια σχόλια με την ε, Μαριάν Χάρκιν. Θα θέλαμε κάποιες μικροαλλαγές ε, σε μερικές συμβαστικές τροπολογίες για να μπορέσουμε να τις υπερψηφίσουμε. Και θα ήθελα επιπλέον να επισημάνω ότι στην παράγραφο 54, όπου γίνεται μια της έκθεσης ε, Omen Reuten, είναι μια μικρή, διατύπωση, μια μικρή αλλαγή στη διατύπωση, αλλά μεγάλη διαφορά στο πώς αντιμετωπίζει κανείς το προσδόκιμο ζωής. Γιατί είναι σαφή η θέση τη ομάδα και φάνηκε και στη συζήτηση τη έκθεση Όμεν Ρόιτεν. Οπότε, αν θέλετε ε, να εμείνετε στη μνήμα τη κυρία Όμεν Ρόιτεν, θα πρέπει να αναφέρετε και την ίδια τη διατύπωση, να μεταφέρετε πιστά την αντίστοιχη παράγραφο της έκθεσης Omen γιατί αυτή η μικρή αλλαγή αλλάζει ουσιαστικά την ουσία. Επίσης, ε, συμφωνώ με τη Μάριον ότι οι δύο επιτροπές έχουν διαφορετικές αρμοδιότητες, οπότε οι εκθέσεις συζητώνται εκ παραλλήλου και ε, ξεχωριστά. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα πρέπει να είναι αντιφατικές. Θα πρέπει να υπάρχει κάποια σύγκληση, ευθυγράμμιση μεταξύ τους, γιατί αν είναι συναφείς εκθέσεις θα ισχυροποιηθεί και η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και έρχομαι εδώ στο θέμα των παραρτημάτων. Ήταν από την αρχή σαφές ότι η, η κρατούσα γνώμη στην ΕΚΟΝ ήταν κατά τη συμπερίληψη των παραρτημάτων. Για πολλού και διάφορου λόγου, όχι λόγω έλλειψη δημοκρατική λογοδοσία. Το αντίθετο, αλλά γιατί μερικά τμήματα του παραρτήματος ήταν μια επίφαση μόνο δημοκρατικής νομιμοποίησης. Εμείς προτιμούμε μια ουσιαστική συζήτηση για το πώς μπορούν να γίνουν πιο δημοκρατικά υπόλογα και το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και Οικονομική Προσανατολισμή. Και ένα από τα σημαντικά θέματα της έκθεσης μου είναι ακριβώς συστάσεις για το μέλλον. Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ πιο επικοδομητικός τρόπος από μια στήρια συζήτηση αν είμαστε υπέρ και κατά του παραρτήματος και τι θα υπάρχει στο παράρτημα. Γιατί είναι πολύ ε, ξύλινες οι κατευθυντήριες γραμμές που περιλαμβάνονται στα παράρτηματα. Και αν θέλουμε συζήτηση με το Συμβούλιο και την Επιτροπή για τι συστάσει αυτέ οικονομική και κοινωνική πολιτική, θα πρέπει οι συστάσει αυτέ να στηρίζονται σε μια εμπεριστατωμένη ανάλυση. Δεν συμφωνώ να έχουμε παραρτήματα που θα προκύπτουν μετά από μια συζήτηση που ο καθένα θα προσθέτει το δικό του. Θα πρέπει να γίνει μια σοβαρή συζήτηση, όχι μόνο μεταξύ μας, αλλά και με το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Και γι' αυτό ακριβώ το λόγο η Επιτροπή ΕΚΟΝ αποφάσισε να βγάλουμε από την έκθεσή μου τα παραρτήματα. Και γι' αυτό ακριβώ το λόγο πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να ασχοληθούμε σήμερα με τα παραρτήματα, γιατί μπορεί να χρησιμοποιηθούν ω επίφαση δημοκρατική νομοποίηση, αλλά δεν συμβάλλουν ουσιαστικά στη συζήτηση για το πόσο μπορεί πραγματικά η όλη διαδικασία να γίνει δημοκρατική και θα μπορούσατε να το αναφέρετε όπως κάνω εγώ στην ε, έκθεση ΕΚΟΝ. Γιατί αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια ουσιαστική συζήτηση για το πώς θα αποκαταστήσουμε κάποια στοιχεία, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε περισσότερο διακυβερνητική μέθοδο παρά κοινοτική. Αυτή η συζήτηση είναι πολύ πιο ουσιαστική από μια συζήτηση μόνο για τα παραρτήματα. Αυτή ήταν η επιχειρηματολογία που ακολούθησε η Επιτροπή ΕΚΟΝ για να αποσύρει από τη συζήτηση τα παραρτήματα. Θέλει άλλος κανείς το λόγο, λέει πρόεδρος. Αν όχι, θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση για τη συμβαστική τροπολογία όμικρον. Πιστεύω ότι η διατύπωση θα δημιουργήσει προβλήματα παραδεκτό. Θα πρέπει να αλλάξουμε τις μνήες, τις εκθέσεις ε, Λοπέ Φοντανιέ και Εστρέλα. Δεν αρκεί μια μνήα του ονόματος έκθεση, πρέπει να είναι πιο ουσιαστική η παραπομπή. Και ελπίζω και ο συγγητή να συμφωνήσει με την αλλαγή στην αιτιολογική σκέψη όμικρων προκειμένου να γίνει τελικά αυτή παραδεκτή, γιατί με τη μορφή που έχει τώρα δεν είναι παραδεκτή. Και του δίνω το λόγο για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Ο κύριος Πριέτο. Ευχαριστώ σε σχέση με τη συμβαστική λύση που αφορά την αιτιολογική ψιόμικρων, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι δεν θα υποβληθεί η σχετική συμβαστική τροπολογία. Θα ψηφίσουμε την αρχική παράγραφο με τις, με τις μεμονωμένες τροπολογίες. Οπότε αυτή η συμβαστική λύση θα αποσυρθεί και θα επανέλθουμε στις μεμονωμένες τροπολογίες για την αιτιολογική σκέψη όμικρον και την αρχική παράγραφό της. Αυτά θα ήθελα να πω στην κυρία Χάρκιν και την Πρόεδρο. Μία διευκρίνηση τώρα. Φαίνεται ότι βρισκόμαστε όλο και πιο κοντά στη συνένεση. Αυτό κατάλαβα από τη συζήτηση γιατί τώρα οριστικοποιούνται οι λεπτές αποχρώσεις των συμβαστικών τροπολογιών. Από τις ε, πολλές συνεδριάσεις που είχαμε με τους σκιώδεις συγητές για να εκπονήσουμε τις συμβαστικές λύσεις, προέκυψε μια πολύ σημαντική γενική συμφωνία, γιατί στις διαπραγματεύσεις των ομάδων εργασίας ο κάθε ευρωβουλευτής εμένει στη θέση του ή στηρίζει τη δική του τροπολογία. Η συμβαστική τροπολογία όμως έχει το χαρακτήρα του συμβιβασμού. Όλοι πρέπει να κάνουμε υποχωρήσεις. Και η έκθεση είναι πολύ σημαντική. Και σε μερικέ παραγράφους έχουμε ιδέες που ενδιαφέρουν περισσότερο τους σοσιαλιστές και παρόλα αυτά υποχωρήσαμε χάρη της Γενικής Συμφωνίας και το ΕΛΚ έκανε το ίδιο σε άλλα σημεία. Δεν θα πρέπει τώρα μια μέρα παραμονές της ψηφοφορίας να εμένει κανείς ή να προσπαθεί να τροποποιήσει ορισμένα πράγματα για να πετύχει να ικανοποιήσει περισσότερο την ομάδα του. Μέχρι στιγμής είχαμε πολύ καλό κλίμα στι διαπραγματεύσεις. Και δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι όλοι κάναμε υποχωρήσεις σε όλες τις συμβαστικές τροπολογίες για να διευκολύνουμε την επίτευξη συνολικής συμφωνία. Τώρα, σε ό,τι αφορά την τροπολογία που ανέφερε ο κύριος Ντεμπάκερ για τις συντάξεις πολύ λεπτό αυτό το θέμα των συντάξεων. Το συζητήσαμε σε δύο εκθέσεις, στην Λευκή Βίβλο, στην Πράσινη Βίβλο, για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και είπαμε να επανέλθουμε σε κοινέ μας θέσεις. Όπως φάνηκαν από τις διάφορες εκθέσεις για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και για την ε, ε, ετήσια επισκόπηση για την ανάπτυξη και για τις ειδικές συστάσεις αναχώρα. Οπότε κύριε Ντεπάκερ, παρακαλώ, μπορεί να μην ε, περιμένατε κάτι τέτοιο, μια ειδική μνήμα, αλλά σας υπενθυμίζω ότι πρόκειται για μια πολύ λεπτή ισορροπία που έχουμε βρει. Και είναι πολύ σημαντικό να διαφυλάξουμε αυτή τη Γενική Συμφωνία και τη λεπτή ισορροπία από το να επιμένουμε ο καθένας σε μία λέξη που θέλει να βάλει να βγάλει. Και συμφωνώ με τον κύριο Ντεμπάκερ ότι η ώψη της Ολομέλειας θα πρέπει να διαμορφώσουμε τις εκθέσεις ώστε να είναι όσο πιο συμπληρωματικές γίνεται. Αλλά δεν θα πρέπει να θεωρείτε τη δική σας έκθεση επιτρεπής εκών ιεραρχικά ανώτερη από την δική μας, της Επιτροπής Απασχόλησης. Και το λέω γιατί η έκθεση Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων αναφέρεται στην αγορά εργασία σε πολλά σημεία. Αναφέρεται στην ανάγκη μεταρρυθμίσεων στον ε, τομέα της εργασίας. Αυτές θα μπορούσαν με βάση τη συσταλτική ερμηνεία και τις αρμοδιότητες να κρυθούν ως μη παραδεκτές. Ακριβώς όμως επειδή θεωρούμε ότι είναι συμπληρωματικές εκθέσεις, το δεχόμαστε. Αλλά ακριβώς επειδή αναζητούμε συμβαστική λύση, θα πρέπει να αποφύγουμε τις περιστάσεις ή τις ε, ιδέες που θα μας ε, εμποδίσουν να καταλήξουμε σε συμβαστική λύση. Επαναλαμβάνω, οι σκιώδεις ηγητές έκαναν πολύ καλή προεργασία και προσπάθησαν πολύ για να καταλήξουμε στη συνένεση. Και οι προτάσεις που έγιναν το πρωί και από τους φιλελεύθερους και από το ΕΛΚ αλλά και από τους πράσινους είναι, όλες οι προτάσεις αυτές είναι λογικές. Οπότε μπορούμε να δεχτούμε ένα ακόμη σημείο να μας να, είναι, να μας λίγο, να μας φίξετε λίγο ακόμη περισσότερο το λουρί. Αλλά όχι παραπέρα. Είμαστε πολύ κοντά στη συμφωνία, παραλαμβάνω, δεν θα πρέπει για μικρολεπτομέρειες να διακινδυνεύσουμε τη συμφωνία για μια πολύ καλή έκθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Καταλαβαίνω πως μετά από την ψηφοφορία στην Επιτροπή θα γίνει και μια συζήτηση του εισηγητή με τις ομάδες ώστε να επαληθευτεί πως δεν υπάρχουν πολλές ε, αντιφάσεις σε σχέση με τα όσα ψηφίστηκαν στην Ολομέλεια. Τώρα, όσον αφορά το περιεχόμενο της έκθεσης του κυρίου Ντιμπάκερ, στην ΕΚΟΝ, είναι αλήθεια ότι δεν το έχουμε εξετάσει όσον αφορά το πεδίο των αρμοδιοτήτων. Αλλά θα γίνει αυτό, διότι ε, η αμοιβαιότης ισχύει και λόγω παραλληλισμού θα πρέπει να το εξετάσουμε εκ του σύνεγγης. Η ναι, και στο κύριο Πριώτο θα ψηφιστεί αύριο και θα πάει στην Ολομέλεια στη Σύνοδο τη 2η του Φεβρουαρίου μαζί με την έκθεση του κυρίου Ντεμπάκερ. Ολοκληρώσαμε την εξέταση αυτού του σημείου και περνάμε στο σημείο 7 όπου θα εξετάσουμε το σχέδιο γνωμοδότησης της ε, προς την Επιτροπή μάλλον Ήτρε. Όχι, διορθώνει η Πρόεδρος. Λοιπόν, εξετάζουμε το σχέδιο έκθεσης. επί το οποίο είμαστε αρμόδιοι επί της ουσίας. Πρόκειται για μια πρόταση οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με του ναυτικού, που τροποποιεί τι οδηγίε 2008-94, 2009-38, 2002-14, 98-59 και 2001-23. Δίνω τώρα λόγο στην εισηγήτριά μας, την κυρία Ροντζούλη, για μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Κυρία εισηγήτρια, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομη. Μετά από 7 χρόνια προτάσεων ε, δημόσιων διαβουλεύσεων, διαφόρων ε, μελετών αντικτύπου, ε, τελικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε, παρουσίασε στις 18 Νοεμβρίου μία πρόταση αναθεώρησης 5 οδηγιών για να βελτιωθούν τα δικαιώματα των ναυτικών που εργάζονται σε πλοία που φέρουν σημαία ε, ενός από τα 28 κράτη-μέλη. Πρόκειται για μια πρόταση που αναμενόταν τον Ιούλιο. Ωστόσο, η Κομισιόν καθυστέρησε και τελικά το παρουσίασε μόνο στους τελευταίους μήνες της θητείας της. Θα ήθελα επίσης να τονίσω πως η Προεδρία η Ελληνική ανακοίνωσε πως δεν θεωρεί ως θέμα προτεραιότητας το εν λόγω θέμα. Ε, όμως θα ήθελα να σας καθησυχάσω ότι εγώ δεσμεύομαι να ολοκληρώσω αυτή την κοινοβουλευτική διαδικασία σε πρώτη ανάγνωση και τον Απρίλιο δηλαδή και ευχαριστώ από τώρα τους συναδέλφους για την προσήλωσή τους και για τη συνεργασία που είμαι βέβαιος, βέβαια ότι θα μου προσφέρουν. Να σας παρουσιάσω εν συντομία την πρόταση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να αναθεωρήσει αυτές τις πέντε οδηγίες για να βελτιώσει τα δικαιώματα των εργαζομένων στον τομέα της ναυτιλίας και να δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης σε ένα κεντρικό τομέα για την ευρωπαϊκή οικονομία. Οι πέντε οδηγίες λόγω είναι η Οδηγία 2008 2008-74 που έχει σχέση με την προστασία των εργαζομένων που σε περίπτωση αφαιρεγγιότητας ε, του εργοδότη. Η Οδηγία 38 του 2009 που αφορά τη δημιουργία μιας επιτροπής επιχείρησης, Ευρωπαϊκής Επιτροπής Επιχείρησης, η Οδηγία 2002-2014 που δημιουργεί ε, γενικό πλαίσιο ενημέρωσης και διαβούλευσης των εργαζομένων και η οδηγία 98 59 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν τις ομαδικές απολύσεις και τέλος την οδηγία 2001-23 σχετικά με τη διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβιβάσεων επιχειρήσεων. Εγώ προσωπικά στηρίζω αυτό το στόχο, αλλά δεν συμμερίζομαι ορισμένα στοιχεία που βρίσκονται στη βάση αυτής της πρότασης. Οι ναυτικοί, αν και ε, εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής ε, των οδηγιών που μόλις σας απαρίθμησα, χαίρουν προστασίας που θεσπίζεται ήδη από τα κράτη-μέλη σε αυτό το τομέα. Δεν νομίζω λοιπόν πως είναι σωστό να κάνουμε λόγο για αποκλεισμό, αλλά καλύτερα θα ήταν να μιλάμε για διαφορετική νομοθεσία. Οι παρατηρήσεις που θέλω να σας ε, απαριθμίσω θα αφορούν ε, την ε, κάθε οδηγία γιατί έτσι είναι πιο απλό. Όσον αφορά την οδηγία σε περίπτωση που αφορά τις περιπτώσεις αφαιρεγγιότητας του εργοδότη. Συμφωνώ εν γέννη με την πρόταση της Κομισιόν. Θεωρώ πως είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί στον εργαζόμενο η δυνατότητα να λαμβάνει τον μισθό του σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν μπορεί να πληρώνει τους εργαζόμενους του και η πρόταση προβλέπει κάθε κράτος μέλος να δημιουργήσει ένα ταμείο εγγυήσεως. Ένα εγγυητικό ταμείο, πολλά κράτη-μέλη ήδη έχουν υιοθετήσει σχετικές εθνικές νομοθεσίες. Για παράδειγμα, στην Ιταλία ε, η Ιταλία ασφαλίζει τους ναυτικούς που βρίσκονται σε τέτοια κατάσταση, δηλαδή φεργιότητα από πλευρά του εργοδότη, ε, μία Προβλέπεται δηλαδή μεταφορά τους ε, στο κοντινότερο αεροδρόμιο και τρεις μήνες αποζημίωσης ε, για αυτούς τους εργαζόμενους. Τώρα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχείρησης. Η πρόταση προβλέπει ότι κάθε επιχείρηση ή ομάδα όμιλος επιχειρήσεων να έχει στο εσωτερικό της μια επιτροπή ε, διαβούλευσης με τους εργαζόμενους. Και σε περίπτωση αυτή πολλές εθνικές νομοθεσίες προβλέπουν ήδη κάποιο τέτοιο σύστημα και χάρη στην παρουσία συνδικαλιστικών εκπροσώπων. Εγώ προτείνω μια ρήτρα επί τη βάση της οποίας σε περίπτωση που ο πρόσωπος ε, των εργαζομένων ε, είναι περιορισμένο σε κάποιο σκάφος και δεν μπορεί να συμμετέχει στην συνδρίαση της Επιτροπής αυτής, ο εργαζότης θα πρέπει να ενημερώσει τον συνδικαλιστικό εκπρόσωπο, έτσι εγγυάται την ενημέρωση και διατηρείται και το δικαίωμα ενημέρωσης του εργαζόμενου και όσον αφορά την 2014 που αφορά την δημιουργία ενός γενικού πλαισίου για την ενημέρωση και τη διαβούλευση με τους εργαζόμενους θα έλεγα όπως και προηγουμένως ότι προβλέπεται η συμμετοχή των εργαζομένων στις, λήψεις, στις αποφάσεις της εταιρείας ε, για τις εταιρείες που έχουν, ε, πάνω, ε, που έχουν 50 εργαζόμενους. Μιλάμε λοιπόν για μια ρήτρα επί τη βάση της οποίας όταν ο εργαζόμενος βρίσκεται πάνω στο πλοίο και δεν μπορεί να συμμετέχει στη διαβούλευση, ο εργοδότης ε, να έχει την υποχρέωση να τον ενημερώσει για κάθε απόφαση που λαμβάνεται στην ε, συνέλευση της Επιτροπής. Τα σημεία 4 και 5 είναι τα πιο επίμαχα. Η οδηγία 98-59 είναι το θέμα που αφορά τις μαζικές απολύσεις, ομαδικές απολύσεις. Προβλέπει λοιπόν η πρόταση ότι ο εργοδότης ο οποίος προτίθεται να προβεί σε ομαδική απόλυση έχει την υποχρέωση να διαβουλευτεί με τους εκπροσώπους των εργαζομένων για να φτάσουν σε κάποια συμφωνία. Εκεί θα πρέπει να συζητηθεί δυνατότητα αποφυγής των απολύσεων ή και να περιορισμός αυτών, να περιορίσουν βέβαια και τις επιπτώσεις τους, ας πούμε κοινωνικά μέτρα, και να προβλέψουν συνοδευτικά μέτρα. Δηλαδή, ο εργοδότη ενημερώνει γραπτό σε την αρμόδια αρχή, επίσης διαβιβάζει αντίγραφο της κοινοποίηση προς του εργαζόμενου που μπορούν να διαβιβάσουν με τη σειρά τους τις δικές τους παρατηρήσεις στις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ε, οι ομαδικές απολύσεις τίθεται δε σε εφαρμογή όχι νωρίτερα από 30 μέρες πριν από την κοινοποίηση. Υπάρχουν ήδη στα κράτη-μέλη νομοθεσίες που προστατεύουν τους εργαζόμενους σε περίπτωση ομαδικών απολύσεων. Η επέκταση λοιπόν, η παράταση της οδηγίας θα δημιουργούσε περαιτέρω γραφειοκρατικό κόστος και διοικητικό κόστος, φόρτο ιδιαίτερα αυτή η περίοδος των 30 ημερών που ονομάζεται και περίοδος προγραμματισμού δεν διαλαμβάνει υπόψη την ιδιαιτερότητα του, ναυτικού, του ναυτιλιακού τομέα και έπειτα ε, οι 30 μέρες μπορεί να οδηγήσουν στην απώλεια ανταγωνιστικότητας. Επιπλέον η άλλη μου παρατήρηση είναι ότι από τη στιγμή που έχει επιτευχθεί συμφωνία με τους κοινωνικούς εταίρους θα πρέπει να περιμένουν άλλες 30 μέρες, πράγμα το οποίο μπορεί να αντιστοιχεί σε αποτυχία των διαπραγματεύσεων και άρα σε ελλειπή προστασία του ίδιου του εργαζόμενου που ε, ίσως ε, σε, μέσα σε αυτές τις 30 μέρες θα μπορεί να το ξανασκεφτεί. Άρα λοιπόν εδώ ή θα πρέπει να μείνουμε στα αυτά, είτε να καταργηθεί αυτή η προθεσμία των 30 ημερών. Τελευταίο σημείο για το, στην περίπτωση μεταβίβασης της ναυτιλιακής επιχείρησης. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η μεταβίβαση επιχείρησης μπορεί να γίνει μετά από πώληση η συμβατική εκχώρηση ή μετά από μια συγχώνευση ανάμεσα σε επιχειρήσεις. Η οδηγία εφαρμόζεται για όλες τις επιχειρήσεις ιδιωτικές ή δημόσιες που ασκούν οικονομική δραστηριότητα. Σε αυτή την περίπτωση οι εργαζόμενοι διατηρούν τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντά τους και απέναντι στον νέο ιδιοκτήτη. Η πρόταση της Κομισιόν δεν μας βρίσκει σύμφωνος για δύο βασικούς λόγους. Όπως έλεγα προηγουμένως, πρόκειται για ένα τομέα ιδιαίτερα διεθνοποιημένο. Τα, οι αλλαγές, οι μεταβιβάσεις ε, ιδιοκτησίας των πλοίων είναι ε, πάρα πολλές, πολυάριθμες και συχνές. Οι εταιρείε θα, αν έπρεπε να σεβαστούν μια πιο αυστηρή νομοθεσία για την μεταβίβαση πλοίων με πιο μεγάλο γραφειοκρατικό φόρτο ε, αλλά και διοικητικό κόστος σίγουρα θα ε, έχαναν απέναντι σε άλλους ε, εξοκοινωτικούς ανταγωνιστές τους. Τώρα, Επίσης, επειδή πρόκειται για κινητές αξίες, για τα πλοία δηλαδή, μπορεί αυτά να είναι γεγραμμένα σε διαφορετικά νιολόγια ε, και είναι πολύ εύκολο να φανταστεί κανείς τις αρνητικές επιπτώσεις στο σε οικονομικό επίπεδο και σε επίπεδο απασχόλησης ε, που προκύπτει από μείωση των ευρωπαϊκών στόλων υπέρ των εξοκοινωτικών στόλων. Έπειτα, οι ναυτικοί που εργάζονται σε κοινοτικά πλοία χαίρουν ε, πάντοτε πνοϊκότερη νομοθεσία. Εάν λοιπόν φύγουν τα κοινοτικά σκάφη προ άλλε σημαίε, θα χαθούν θέσει εργασία αλλά και ναυτικοί, οι οποίοι για να μην χάσουν τη δουλειά τους θα αναγκαστούν να εργαστούν χωρίς την προστασία της ε, κοινοτικής νομοθεσίας, εκτός που θα υποχρεωθούν να μεταφερθούν και οι ίδιοι. Ε, Άρα λοιπόν η οδηγία για τη μεταβίβαση των επιχειρήσεων θα πρέπει να αλλάξει για τον τομέα της ναυτιλίας. Μου ζητήσατε να συντομεύω, οπότε ε, θα σταματήσω σε αυτά που είπα μέχρι τώρα. Τώρα, αν οι συνάδελφοι έχουν ερωτήσει, ε, να κλείσω αργότερα. Ευχαριστώ. Euh. Σας ευχαριστώ για την λεπτομερή ανάπτυξη του θέματος της εκθέσεώς σας. Το λόγο δίνω πάλι στον κύριο Ντεμπάκερ. Άλλος επιθυμεί κανείς να παρέμβει. Μόνο εσείς. Καλά. Όχι κυρία Χάρκιν, όχι, όχι. Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Πρώτα ο κύριος, Ντεμπάκερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ με την ευκαιρία και την ε, ίδια την εισηγήτρια. Πρόκειται για μια εξαιρετικά χρήσιμη πρόταση. Η έκθεση είναι πολύ λογική και μας δίνει μια καλή επισκόπηση της κατάστασης των προσώπων αυτών. Δεν είμαι απαραίτητα θερμός υποστηρικτής των προτάσεων της Κομισιόν. Και νομίζω ότι ε, η συγγήτρια επαναφέρει την Κομισιόν σε κάτι πιο λογικό. Αντιλαμβάνομαι ότι η Κομισιόν θέλει να προσαρμόσει την νομοθεσία των ναυτεργατών για να γίνουν οι θέσεις αυτές πιο ελκυστικές και για τους νέους, να ενισχυθεί ο τομέας, διότι υπάρχει πτώση και άρα να γίνει κάποια προσπάθεια να γίνει ο τομέας ελκυστικότερος. Όμως δεν είμαι βέβαιος ότι η Κομισιόν έχει επιλέξει τη σωστή προσέγγιση. Ορισμένους λόγους ανέπτυξε ήδη η συγγήτρια. Οι ναυτεργάτες δεν έχουν την ίδια, το ίδιο καθεστώς με αυτούς που εργάζονται ε, σε χερσαίες επιχειρήσεις. Είναι θέμα και κοινωνικών ασφαλίσεων. Έχουν όμως και ορισμένα πρακτικά προβλήματα τα οποία θα προκύψουν εάν εφαρμοστεί ισότιμα η νομοθεσία στους ναυτεργάτες όπως ε, σε αυτούς που εργάζονται στην ξηρά. Υπάρχουν για τους ναυτεργάτες ιδιαίτερα καθεστώτα όπως ο IMO, ο οργανισμός δηλαδή ναυτιλίας, αλλά το διεθνές επίπεδο δεν είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί ο τομέας είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικός. Είναι πολύ εύκολο να μετακινηθεί το πλοίο από ένα λιμάνι σε άλλο και βεβαίω το ίδιο, όχι το ίδιο εύκολο, αλλά πάντως είναι εύκολο να μετακινηθεί και από μία σημαία σε άλλη. Η 2001-23 οδηγία, έχω και εγώ τη γνώμη εδώ, εάν αναγκάσουμε τους, εργο, τους εργοδότες να προσλάβουν τα ίδια άτομα, αυτό θα έχει ε, τελικώς ε, τα αντίθετα αποτελέσματα, διότι εφόσον αλλάζει ο κύριος του πλοίου, αλλάζει και η σημαία και ενδέχεται το πλήρωμα να βρεθεί σε δυσκολότερη θέση. Αυτά τα σχόλια έχω για την ώρα. Κατά τα άλλα συμφωνώ με την εισηγήτρια και ίσως ε, μπορέσουμε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με τον επικοδομητικό αυτό τρόπο. Ευχαριστώ. Μιλούμε για περίπου μισό εκατομμύριο ε, ναυτεργάτες και ψαράδες. Και βεβαίω ο ευρωπαϊκός στόλος είναι το 20% του παγκόσμιου στόλου. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για ε, το ναυτεργατικό επάγγελμα. Συζήτηση που συνεχίζεται και έχει ως στόχο να βρει τρόπο να, βελτιωθούν, να βελτιωθεί η κατάσταση των ε, ναυτικών. Και είχαν όλοι την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους για το μέλλον του τομέα. Η βελτίωση των δικαιωμάτων των εργαζόμενων σε όλους τους τομείς είναι ένας από τους στόχους για την δημιουργία της κοινωνικής Ευρώπης. Και στους διάφορους τομείς βεβαίω είναι αυτό απαραίτητο. Ως εκπρόσωποι των λαών οφείλουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα συνεχίσουμε να κατανοούμε τις προκλήσεις των ενδιαφέρων τομέων και τις επιπτώσεις τους εργαζόμενους. Ο, τομέας, ο ναυτιλιακός τομέας είναι ιδιαίτερος. Πρέπει να γίνει σχετική ανάλυση με τρόπο που να μην έχει αρνητικές επιπτώσεις στις συνθήκες εργασίας των, των ναυτικών. Πρέπει να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα υπέρ των εργαζόμενων. Αυτό είναι απαραίτητο έτσι ώστε οι συνθήκες των εργαζόμενων σε κάθε τομέα να βελτιωθούν και οι τομείς να προσελκύσουν εργαζόμενους, τομείς οι οποίοι ενδεχομένως δεν θεωρούνται πλέον ελκυστικοί. Και βέβαια ο, το ναυτιλιακός τομέας είναι ένα σχετικό παράδειγμα. Από όλα τα έγγραφα και άλλες εκθέσεις που έχουν υποβληθεί προκύπτει το συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν επαρκεί πληρώματα με τις απαραίτητες δεξιότητες για να επανδρώσουν τα ευρωπαϊκά πλοία. Είναι σημαντικές οι προκλήσεις λοιπόν και πρέπει κανείς να μην λησμονεί ότι υπάρχουν και βελτιώσεις που έχουν επιτευχθεί ως αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων και του διαλόγου. Η διαδικασία στη βάση διαβουλεύσεων με τους ενδιαφερομένους έχει φωτίσει ορισμένα θέματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη από τις πιο σημαντικές εγγυήσεις που δίνονται στους εργαζόμενους στον αυτιλιακό τομέα προκύπτει από την ILO Maritime Convention και που έχει τεθεί σε ισχύ και που προσφέρει, εγγυάται ορισμένα δικαιώματα. Η περαιτέρω βελτίωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων πρέπει να προκύψει μέσα από διαρκή διάλογο μεταξύ εργοδοσίας και των επικεφαλής των εργατικών συνδικάτων έτσι ώστε να υπάρξει ισορροπία μεταξύ των συμφέροντων των δύο μερών. Η συζήτηση που διεξάγουμε τώρα για τις τροπολογίες ασφαλώς προσφέρει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση καθώς και βέβαια μια ζωντανή συζήτηση. Η Κομισιόν έχει λάβει μια ενεργητική προσέγγιση στην πρόταση που έχει κάνει. Όμως η έκθεση της Κομισιόν δείχνει ότι υπάρχουν διάφορες επιλογές πολιτικής για την αντιμετώπιση των θεμάτων. Εν τέλει τα δικαιώματα των εργαζομένων πρέπει να προστατεύονται και να είναι εξασφαλισμένα. Όμως η προσέγγιση πρέπει να τέτοια που να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες όλων των μερών. Γιατί έχουμε απέναντί μας δύο διαφορετικές θέσεις. Αφενός την Κομισιόν που βγαίνει προς μια κατεύθυνση και την εισηγήτρια που πηγαίνει προς αλλού. Θα είναι λοιπόν σημαντική και ενδιαφέρουσα η πρόκληση. Σε ό,τι αφορά ορισμένες προτάσεις μπορεί να θεωρήσει κανείς ότι οι τεχνολογικές πρόοδοι θα βοηθήσουν έτσι ώστε να προσελκυστούν περισσότεροι εργαζόμενοι στον τομέα. Αυτό ίσως είναι σημαντικό για την προσέγγιση που λαμβάνει η, η Οι οδηγίες που θα ψηφιστούν πρέπει να, είναι, να λάβουν υπόψη τα, τα συμφέροντα των εργαζομένων. Βέβαια, πρέπει να έχει κανείς και υπόψη την διάκριση μεταξύ χερσαίων εργαζόμενων και των ναυτικών από την άλλη μεριά. Να μην γίνει καμιά αλλαγή που να βλάψει τον τομέα. Αναμένω με ενδιαφέρον λοιπόν την συνεργασία και με την εισηγήτρια αλλά και με τους άλλους κοιόδης εισηγητές για τον φάκελο αυτό. Ευχαριστώ. Θέλει άλλος κανείς το λόγο. Όχι, οπότε να ρωτήσω αν υπάρχει εδώ εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θέλει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή Απασχόληση και ιδιαίτερα την εισηγητρία γιατί αντέδρασε άμεσα στην πρόταση του Νοεμβρίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κατέρτησε έκθεση. Όπως είπαν οι προλαλήσαντες, μία σύντομη υπενθύμηση των βασικών στόχων της πρότασης βελτίωση των συνθηκών ζωής και εργασίας των ναυτικών, χορηγώντας τους τα ίδια δικαιώματα με αυτά που έχουν και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι, αυτοί που εργάζονται στην ξηρά. Ε, καταργούμε την ανομαλία αυτή της εξαίρεσης ε, των ναυτικών από πολλές ευρωπαϊκές οδηγίες που αφορούν τα δικαιώματα των εργαζομένων. Ήταν τελείως παράλογη αυτή η εξαίρεση. Επίσης προσπαθούμε να διαμορφώσουμε συνθήκες ισότιμου ανταγωνισμού στην ναυτιλία, στον ναυτιλιακό κλάδο στην Ευρώπη. Γιατί θα πρέπει και οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις αλλιές να υπόκειται στις ίδιες ανάγκες ισότιμου ανταγωνισμού. Λαμβάνουμε υπόψη όπως και τις ιδιαιτερότητες του ναυτιλιακού τομέα στην Ευρώπη. Γιατί υφίσταται πολύ μεγάλο ανταγωνισμό από ε, τρίτες χώρες ε, εξαιτίας της αλλαγής ε, σημαίας και γι' αυτό χρειάστηκε να κάνουμε κάποιες αλλαγές στην πρόταση για να λάβουμε υπόψη αυτά τα θέματα αλλά και το κόστος. Όπως είπε η τελευταία ομιλήτρια, οργανώσαμε εκτεταμένες διαβουλεύσεις και με τους κοινωνικούς εταίρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Περιμένουμε γενική υποστήριξη για την προσέγγιση μας και ε, ευελπιστώ ότι θα υπάρχει και συνέχεια σε αυτή την υποστήριξη. Ελπίζω να μην αποδυναμωθούν κάποιες διατάξεις για να μην έχουμε παλινδρόμηση σε σχέση με την παρούσα κατάσταση. Ακόμη και στα κράτη-μέλη που ήδη επέλεξαν να συμπεριλάβουν τους ναυτικούς στο πεδίο εφαρμογή των ευρωπαϊκών οδηγιών για τα εργασιακά δικαιώματα. Τώρα, κάποιες μεμονωμένες παρατηρήσεις ε, για τις ε, απόψεις που ακούσαμε. Η σχετική συνθήκη του ΔΟΕ, της ΔΟΕ, της Διεθνής Οργάνωσης Εργασίας για, για την αυτιλία. Οι συνθήκε αυτές περιλαμβάνουν ελάχιστου κανόνες και προδιαγραφέ για τις συνθήκε ζωής και εργασίας των ναυτικών. Για παράδειγμα, δικαίωμα ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, δικαίωμα κοινωνικής προστασίας, κοινωνική ασφάλεια και προβλέπει το δικαίωμα κατάρτισης και επιμόρφωσης των εργαζομένων ή δικαιώματα σε περίπτωση μαζικών απολύσεων ή μεταφοράς επιχείρησης και σε θέματα μεταφοράς επιχειρήσεων θα ήταν κρίμα να αποκλείονται οι ναυτικοί από οποιοδήποτε δικαίωμα ενημέρωσης ή προηγούμενης διαβούλευσης. Θέλουμε λοιπόν να, να προσπίσουμε θεμελιώδη δικαιώματα των ναυτικών και σε περίπτωση μεταβίβασης επιχειρήσεων. Σε ό,τι αφορά το θέμα της Επιτροπής Επιχείρησης, Ευρωπαϊκής Επιτροπής Επιχείρησης. Θεωρήσαμε ότι υπάρχουν σύγχρονα και σχετικά φθηνά μέσα για καλύτερη ενημέρωση και επικοινωνία και κρίμα θα ήταν και πάλι να αποκλείσουμε τους ναυτικούς από πρόσκληση και για συμμετοχή σε ενημερωτικές συνεδριάσεις. Γιατί τους άλλως τέτοιες σπάνια γίνονται και πολύ πιο σπάνια προσκαλούνται οι ναυτικοί. Και συνήθως ε, είναι έκτακτες αυτές οι συνεδριάσεις. Δεν θέλουμε λοιπόν να έχουμε επαναχώρηση σε σχέση με το γενικό δικαίωμα ενημέρωσης και διαβούλευσης ε, που προβλέπει η οδηγία του 2002 και δεν θέλουμε επαναχώρηση ή αποδυνάμωση της προστασίας που χορηγεί η οδηγία, ιδιαίτερα στο θέμα της, του επίπεδου ισοδύναμης προστασίας. Σε ό,τι αφορά την οδηγία για τις α, ε, συλλογικές απολύσεις, δεν θέλουμε να δημιουργηθεί μια έλλειψη ασφάλειας δικαίου κατά την εφαρμογή διαφορετικών νομοθεσιών σε ό,τι αφορά την, τις διατάξεις για τις μαζικές απολύσεις. Και σε ό,τι αφορά το σχόλιο της ηγήτριας, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η πρόταση ήδη προβλέπει τη δυνατότητα κατάργησης της περίοδου κοινοποίησης σε περίπτωση πώλησης πλοίου ή σε περίπτωση που πρόκειται για μικρομεσαία επιχείρηση. Λάβαμε δηλαδή υπόψη τον παράγοντα κόστος ή διοικητικές διατυπώσεις. Αυτά και είμαι στη διάθεση της ηγήτριας για περαιτέρω διευκρινήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία εισηγήτρια, έχει το λόγο. Έχετε να σχολιάσετε αυτά που είπε ο κ. Ντεμπέκερ και άλλοι. Ε, Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όχι, ε, δεν έχω να κάνω ακριβώς απάντηση αυτή καθ' γιατί θα συνεργαστούμε έτσι και αλλιώς εργότερα. Εγώ ε, ακούσα τις παρατηρήσεις των συναδέλφων και της Κομισιόν και έχω παρουσιάσει κάποιες αλλαγές σε σχέση με την πρόταση της Κομισιόν που κατά τη γνώμη μου δεν λάμβανε υπόψη κάποιες πραγματικότητες του ναυτικού επαγγελματικού κλάδου και κυρίως τη λειτουργία του τομέα των θαλάσσιων μεταφορών. Η ανάλυση για να απαντήσω στην ε, συνάδελφο Μπαλντακίνο που διάβαζε Αναλύσεις έχουν γίνει έως και υπερβολικές. Ε, περιμέναμε 7 χρόνια ολόκληρα για να λάβουμε αυτή την πρόταση δεν θα ήθελα ούτε να κατευθυνθώ προς μια τελείως διαφορετική κατεύθυνση από αυτή τη Κομισιόν, γιατί ε, αν έπρεπε να ακολουθήσω εντελώς διαφορετική κατεύθυνση, θα ζητούσα και θα απέκλεια τους ναυτικούς και από τις πέντε ε, ε, οδηγίες. Και δεν έκανα τέτοιο είδο πρόταση. Και αυτό γιατί η πρόταση της Κομισιόν δεν ακολουθεί την ε, κατεύθυνση της ανάπτυξης και της ε, ανάκαμψης, ε, πράγμα το οποίο αποζητούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση που πλήττεται από εξαιρετικά υψηλά ποσοστά ανεργίας. θέλω να βρούμε μια ενισορροπία ανάμεσα στα δικαιώματα των εργαζόμενων αλλά και των ασφάλεια δικαίου για όλους τους φορείς του κλάδου. Να δώσουμε δηλαδή στους ε, ε, ναυτικούς την καλύτερη δυνατή ε, νομική κάλυψη, σε αυτό συμφωνούμε όλοι, αλλά και να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την ανταγωνιστικότητά μας που την έχει αυτός ο τόσο ιδιαίτερος τομέας και που καθημερινά απασχολεί, όπως θυμήσατε, 500.000 ναυτικούς. Κλείνω λέγοντας και θυμίζοντας ότι έχετε τη δυνατότητα να υποβάλλετε τροπολογίες μέχρι τις 27 Ιανουαρίου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Συγγέντρια. Να σας θυμίσω ότι για αυτό το κείμενο είμαστε σε διαδικασία συναπόφασης και ότι η ελληνική προεδρία που ωστόσο θεωρεί το θέμα των ναυτικών μεταφορών, των θαλάσσιων μεταφορών προτεραιότητά της, ε, θεωρεί πως αυτό το κείμενο δεν είναι προτεραιότητά της. Και άρα λοιπόν γνωρίζουμε πως θα κλείσουμε αυτή τη θητεία με απλά και μόνο μια πρώτη ανάγνωση από πλευρά του Ευρωκοινοβουλίου. Οι προτάσεις της συζυγήτριας ε, τροποποιούν σε πολλά σημεία την πρόταση που μας υπέβαλε ο Επίτροπος του για να ε, βγουν οι ναυτικοί από αυτή την ιδιαιτερότητα ε, όσον αφορά τα εργατικά τους δικαιώματα και από αυτό το πνεύμα θα δούμε λοιπόν αυτές τις προτάσεις και θα καταθέσουμε τροπολογίες με ψηφιακή υπογραφή μέχρι τις 27 ή Ιανουαρίου το μεσημέρι στις 12. Θα εξετάσουμε τις τροπολογίες αυτές στις 12 και 13 Μαρτίου, συμβιβαστικές 17 ε, Μαρτίου και ψηφοφορία στις 18 και μετά θα πάμε στην Ολομέλεια άμεσα, στη δεύτερη Ολομέλεια του Απριλίου για την πρώτη ανάγνωση. Ολοκληρώθηκε έτσι η εξέταση αυτού του σημείου και περνάμε στο σημείο 8 όπου θα δώσω το λόγο στον Τζάμπα Όρη για να μας παρουσιάσει το σχέδιο προσωρινής έκθεσης για την απόφαση του Συμβουλίου σε σχέση με τη τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφή για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Έχετε το λόγο κύριε Σιγητά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μπορούσαμε να πούμε με βεβαιότητα ότι η αλλαγή αυτή είναι τεχνικού χαρακτήρα. Αφορά την Τριμερή Κοινωνική Σύνοδο Κορυφής, που είναι πια θεσμός και προηγείται της διασκέψης κορυφής της Άνοιξης και του Φθινοπόρου. Έχουν υποβληθεί οι και οι κοινωνικοί εταίροι συμφωνούν με την προσπάθεια αυτή. Πριν συντάξω τις τροπολογίες, είχα συζητήσει και με την Business Europe και την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων και με άλλους εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων και διαπιστώνω ότι όλοι είναι ικανοποιημένοι με το ισχύον σύστημα. Αυτό που τους ενδιαφέρει κυρίως είναι στενότεροι δεσμοί με τους ηθήνοντες και αρμοδίους λήψης αποφάσεων. Αυτή είναι μια πολύ εύλογη απέτηση και λογική. Θεμητή. Άλλωστε αναφέρθηκε και από το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι αυτοί οι τριμερείς, αυτές οι τριμερείς κοινωνικές σύνοδοι κορυφής θεσπίστηκαν με σκοπό την ενημέρωση του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη θέση των κοινωνικών εταίρων. Κατέθεσα μερικές τροπολογίες που λαμβάνουν υπόψη τις προσδοκίες και απαιτήσεις των κοινωνικών εταίρων και τόνισα σε αυτές ότι θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι οι κοινωνικοί εταίροι στέλνουν ε, στην Τριμερή Κοινωνική Σύνοδο Κορυφής έγκυρους εκπροσώπους τους προκειμένου να διαμηνηθεί από αυτές τις συνόδους κορυφής η γνώμη των κοινωνικών εταίρων προς το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, διαπιστώνεται η ανάγκη να υπογραμμίσουμε ότι οι οργανώσεις που εκπροσωπούν διάφορους τομείς καλό θα ήταν να συνεννοούνται και να καταλήγουν ε, σε διακλαδικές ε, κοινέ θέσεις ώστε να έχει μεγαλύτερο σθένος το μήνυμα που θα στείλουν οι κοινωνικοί εταίροι και άρα η μεγαλύτερη βαρύτητα και πιθανότητα να ληφθεί υπόψη από το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι σημαντικό οι θύνοντες ε, πολιτικοί που χαράζουν και λαμβάνουν τις αποφάσεις να λαμβάνουν υπόψη τις θέσεις των κοινωνικών εταίρων. Είμαστε ικανοποιημένοι με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θεωρώ ότι καλό θα ήταν με τις τροπολογίες ε, να συμπληρωθούν ε, ορισμένα σημεία που λείπουν. Αυτά. Και κάτι που ξέχασα για το χρονοδιάγραμμα. Το χρονοδιάγραμμα που προτείνει η Γραμματεία. Ευελπιστώ ότι θα τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμά μας. Το Ερεινό Συμβούλιο έχει προγραμματιστεί για την 10η Μαρτίου ή την εβδομάδα που ξεκινάει στις 10 Μαρτίου αρκεί να υποβληθούν ε, ελάχιστες ή καθόλου τροπολογίες. Δεν είναι πάντως σίγουρο. ότι θα καταφέρουμε να διεκπαιρεώσουμε το έργο μας μέχρι την Ολομέλεια του Μαρτίου. Η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών Λίγη στις 28 Φεβρουαρίου. Ελπίζω να μπορέσουμε να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα που πρότεινε η Γραμματεία. Αυτό θα το καταφέρουμε αν περιοριστούμε περιορίσουμε στο ελάχιστο τον ε, αριθμό των νέων τροπολογιών. Αν οι συνάδελφοι συμφωνούν με τις προτάσεις μου και δεν υποβάλλουν τροπολογίες, θα έχουμε πολύ μεγάλες πιθανότητες να ακολουθήσουμε το χρονοδιάγραμμα. Αυτά. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα, όπως καταλάβατε, με την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ κυρία Παλατσίνο και ο κύριος Δεμπάκερ. Η κυρία Μπαλτακίνο. Η Μπαλτατσίνο. Ευχαριστώ. Χαιρετίζω την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο κοινωνικός διάλογος θα πρέπει να διατηρηθεί δεδομένων των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε σε θέματα ανάπτυξης και απασχόλησης. Η ανάπτυξη και απασχόληση και η, θεμα, θεματολογία της τριμερής κοινωνικής συνόδου κορυφής είναι απαραίτητα θέματα για να αντιμετωπιστεί η σοβούσα οικονομική και κοινωνική κρίση. Η ανάπτυξη και η απασχόληση είναι οι παράγοντες που θα μας επιτρέψουν να εξέλθουμε από την κρίση. Πολλά δε μάλλον που έχουν εφαρμοστεί δρακόντια μέτρα λιτότητας τα τελευταία χρόνια. Σε μια ραγδαία μεταβαλλόμενη οικονομία και με πολλούς τομείς που θα πρέπει να ανακάμψουν μετά την οικονομική κρίση και με τα υψηλά επίπεδα ανεργίας θα πρέπει να αποφύγουμε τον κοινωνικό αποκλεισμό και φυσικά την γενίκευση των επισφαλών θέσεων απασχόλησης. Θα πρέπει σίγουρα να βελτιώσουμε, να ενισχύσουμε την κοινωνική διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γι' αυτό και θα πρέπει να συμπεριλάβουμε στη συζητήση όλους τους κοινωνικούς εταίρους. Είναι αδιανόητο να έχουμε ανάπτυξη και ε, απασχόληση χωρίς εκτενείς διαβουλεύσεις με όλους τους κοινωνικούς εταίρους. Γιατί αυτή είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας ε, και φυσικά αυτοί εφαρμόζουν τις ε, πολιτικές στην πράξη, οι εργοζόμενοι και οι εργοδότες και γι' αυτό η συμμετοχή τους στις διαβουλεύσεις είναι απαραίτητη. Επίσης θεωρώ ότι η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής εμένει στη σωστή πρακτική των δύο κοινωνικών ε, συνόδων κορυφής και αναφέρει και τη στρατηγική του 2020. Χαίρομαι και για την διάμεση αναθεώρηση που προτείνεται, που θα περιέχει συστάσεις. Προσβλέπω στη συνέχεια των συζητήσεων, σε συνεργασία, γιατί είναι θέματα που βρίσκονται στην καρδιά των ευρωπαϊκών πολιτικών. Ευχαριστώ. Φίλιπ Ντεμπάκερ, θέλει άλλος κανείς μετά από εκείνο το λόγο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά πρώτα ο Φίλιπ Ντεμπάκερ. Ευχαριστώ. Εκπροσωπώ εδώ τη Μαριάν Χάρκιν που χρειάστηκε να φύγει και μου ζήτησε να διαβάσω μια σύντομη δήλωσή τη. Η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λέει κυρία Χάρκιν είναι σωστή. Λαμβάνει υπόψη τη ε, θετική συνεδρίαση τη συμμετοχή των τριών διαδοχικών προεδριών στη συζήτηση και παρόλο που δεν απαιτεί νομική βάση, ε, καλό θα είναι να συνεχιστεί αυτή η παράδοση. Η Τριμερής Κοινωνική Σύνοδος Κορυφής ε, ουσιαστικά συνεκλήθη δύο φορές το χρόνο, αν και νομικά απαιτούνταν μόνο η άπαξ ε, σύγκλησή της. Αλλά προτείνουμε να συνεχιστεί αυτή η εξάμηνη τριμερής σύνοδος κορυφής, δηλαδή δύο φορές το χρόνο είναι υπέρ και της έκθεσης όρη η κυρία Χάρκιν. Ευχαριστώ και τώρα να δώσω το λόγο στον Ζων Πολ Τχικάχ, εκ μέρους Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Όρη και τους υπόλοιπους ευρωβουλευτές που έλαβαν το λόγο. Όπως είπε ο κύριος Όρη, πρόκειται για μια τεχνική ουσιαστικά αναθεώρηση που χρειάστηκε να υποβάλουμε για να προσαρμόσουμε τις δομές της τρίμερους ε, κοινωνικής συνόδου κορυφής που υπάρχει από το 2003 στη συνθήκη της Λισαβόνας και στη δημιουργία της νέας θέσης του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου καθώς και στην ε, θέσπιση της στρατηγικής Ευρώπης 2020 που αντικατέστησε την προηγούμενη στρατηγική της Λισαβόνας. Οπότε στόχος της πρότασης είναι να γίνουν κάποιες τεχνικές αλλαγές. Έχουμε όμως πρόβλημα με το χρονοδιάγραμμα που σχετίζεται με τη νομική βάση της πρότασης. Η πρόταση υπευλήθη με βάση το άρθρο 352 που προβλέπει ομοφωνία στο Συμβούλιο με σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με συνένεση. Και προσφύγαμε στο άρθρο 352 γιατί η προηγούμενη νομική βάση της απόφασης καταργήθηκε με τη θέση ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας. Οπότε ήταν απαραίτητο να χρησιμοποιήσουμε μια νομική βάση που για μερικές χώρες μέλη θα καταστήσει πιο χρονοβόρα τη διαδικασία έγκρισης. Γιατί απαιτείται εθνική κοινοβουλευτική διαδικασία για την έγκριση απόφαση σε ορισμένα κράτη-μέλη. Κατά την προετοιμασία ε, για την εκπόνηση της πρώτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής είχαμε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους. Εξάλλου η πρότασή μας στηρίζεται στην μακροχρόνια πια πρακτική που εφαρμόζουμε και ε, άτυπα προσαρμόσαμε αυτές τις τριμερείς κοινωνικές συνόδους κορυφής ε, στο ρόλο του Πρόεδρου Βαν Ρομπόι ως Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και για να εξασφαλίσουμε μια πιο ισορροπημένη κατανομή μεταξύ των συμμετεχόντων στην τριμερή αυτή διάσκεψη κορυφής. Ήταν πολύ ρεαλιστική λοιπόν η πρόταση και είμαστε πρόθυμοι να λάβουμε υπόψη και τη συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πάντως και με το Συμβούλιο και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσπαθήσαμε να υιοθετήσουμε μια τεχνική προσέγγιση δεν πρόκειται να επιλύσουμε όλα τα προβλήματα διαχείρισης, διακυβέρνησης που υπάρχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έπρεπε όμως να λάβουμε μια τεχνική απόφαση για μια αναθεώρηση που καλό θα ήταν να εγκριθεί σε έφθετο χρόνο. Άλλωστε αυτός είναι και στόχος της ελληνικής προεδρίας με την οποία συνεργαζόμαστε στενά. Στόχος είναι να γίνει έγκριση ε, με συμφωνία επί της αρχής ε, πολιτικό επίπεδο στο Συμβούλιο Κοινωνικών Υποθέσεων του Μαρτίου. Οπότε δεν ξεχνούμε το χρονοδιάγραμμα. Βέβαια θα λάβουμε υπόψη και τις τροπολογίες όταν τις εκπονήσετε και τις υποβάλλετε. Θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι τροπολογίες που θα υποβληθούν για την απόφαση αυτή και είναι κυρίαρχο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κρίνει πόσε θα υποβάλει και ποιε θα λάβει υπόψη. Τώρα, ε, στις διάφορες συνεδριάσεις, στις διάφορες εκθέσεις και στα διάφορα ευρωπαϊκά συμβούλια τονίζουμε την ανάγκη βελτίωσης του κοινωνικού διαλόγου. Και τώρα, στο τέλο τη κοινοβουλευτική θητεία και τέσσερα χρόνια μετά τη θέση ισχύ της Διεθήκης Λισαβόνας, βλέπουμε μια πρόταση που μας διαβεβαιώνεται ότι είναι τεχνικής φύσης, απλώς προσθέτει τον κύριο Βαν Ρομπόη αντικαθιστώντας τον πρόεδρο άλλου συμβουλίου και προσαρμόζεται την πρόταση στην συνθήκη της Λισαβόνας και την Ευρώπη του 2020. Μα αν είναι απλώς γραφειοκρατικό το έργο, δεν έπρεπε να περιμένετε τόσα χρόνια για να μας κάνετε μια τεχνική πρόταση και να κάνετε μια τέτοια τεχνική πρόταση χωρίς καν να μπαίνετε στον κόπο να ρωτάτε αν ε, το Κοινοβούλιο έχει να πει κάτι. Πραγματικά είναι παράλογο αυτό. Εντάξει, δεν πρόκειται να κάνουμε επανάσταση με ένα κείμενο που έχει χαρακτηριστεί τεχνικό και δεδομένη στις πίεση χρονοδιαγράμματος που αντιμετωπίζουμε και θα φροντίσουμε να συμφωνήσουμε με το Συμβούλιο πριν το τέλος της κοινοβουλευτικής θητείας. Δεν είμαι καν σκιωδησηγήτρια για το θέμα αυτό. Καθήνα στο σκιωδησηγητή τη διακριτική ευχέρεια για το αν θα θέσει αυτό το θέμα. Μία μικρή θέση έστω και παρατηρητή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πού είναι το δύσκολο θα μπορούσαμε να το ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κρίνει ε, τη σοφία της ε, αν είναι χρήσιμη η παρουσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο κοινωνικό διάλογο. Μπορεί βέβαια η ΕΚΤ να πει ότι δεν έχει θέση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί θα υποβαθμιστεί έτσι η ποιότητα του κοινωνικού διαλόγου. Εν πάση περιπτώσει, για να δώσουμε ένα πιο πολιτικό και δυναμικό χαρακτήρα στη συζήτηση, υπάρχει και το θέμα της διακυβέρνηση, τη οικονομική και Νομισματικής ε, Ένωσης, που ανακύπτει ως θέμα και που δεν είναι καθόλου τεχνικό. Θα, πρέ... θα σας πρότεινα στα πλαίσια της εφαρμογής του άρθρου 81 που μόλις θέθηκε σε ισχύ με τη νέα μορφή, θα πρότεινα παράλληλα με τη διαδικασία έγκρισης consent που θα χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά με την έκθεση του κυριορή να μπορέσουμε όπως προβλέπει η νέα εκδοχή του άρθρου 81 να εφαρμόσουμε εκ, παραλέλ, παραλίλου μία διαδικασία ψηφίσματος με συζήτηση για να μπορέσουμε να κάνουμε μία πολιτική ανάλυση όλων αυτών των θέμα, θεμάτων που αναφέρονται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου εδώ και πολλά χρόνια. Και αυτή η ιδιαίτερα τεχνική πρόταση που έγινε εδώ αναφέρεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Ιουνίου του 2013 για την κοινωνική διάσταση της ΟΝΕ και στην ανακοίνωση του 2013 για την κοινωνική διάσταση της ΟΝΕ. Από ό,τι ξέρω και τα δύο αυτά κείμενα δεν είναι διόλου Πιστεύω, πιστεύω λοιπόν και ελπίζω πως ο εισηγητής ε, θα δει ε, την πρόταση αυτή και θα μπορέσουμε έτσι να έχουμε με μια πρόταση ψηφίσματος που θα μας επιτρέψει να θίξουμε τα πιο πολιτική φύσης θέματα, ελπίζοντας πως θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε κάποια συμφωνία μεταξύ μας επ' αυτού. Και θα ξαναδώσω τώρα το λόγο στον εισηγητή για να κλείσουμε τη συζήτηση για το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ. Εγώ ξεκίνησα την εργασία αυτή με εξαιρετικά ανοιχτό μυαλό. Όντως η Κομισιόν υπέβαλε μια τεχνική φύσης πρόταση και από αυτού ρωτούν τη γνώμη μας και τη συμβολή μας. Εγώ απευθύνθηκα στους κοινωνικούς εταίρους και τελικά οι κοινωνικοί εταίροι ομόφωνα είπαν ότι στην πράξη πρόκειται για την παγίωση πρακτικών που ήδη έχουν καθιερωθεί ε, στις προηγούμενες κοινωνικές ε, συνόδους κορυφής. Δεν πίστευα ότι έπρεπε να εξετάσουμε εις βάθος το θέμα, γιατί ακριβώς οι κοινωνικοί εταίροι φαίνεται να συμφωνούσαν. υπήρχε ήδη συμφωνία δηλαδή θεώρησα. Τώρα το Κοινοβούλιο θέλει να φέρει την συζήτηση αυτή σε πολιτικό επίπεδο, αυτό είναι άλλο ζήτημα. Ε, πάντως είναι μια πρόταση που έρχεται έτσι, ως τελευταία στιγμή και πρέπει να το συζητήσω και με τους άλλους συναδέλφους. Εγώ δεν είμαι κατά του να μιλήσουμε και για πολιτικά θέματα, γιατί αυτή είναι η δική μας δουλειά. Αν λοιπόν είναι προς όφελός μας, θα πρέπει να κάνουμε να και την πολιτική συζήτηση για το θέμα αυτό, αλλά μέχρι στιγμή. υπήρξαν και δεσμεύσει, αλλά πιστεύω πως μπορούμε να το συζητήσουμε ε, μεταξύ μας. Τώρα όσον αφορά την ε, ίδια την πρόταση, Νομίζω πως δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα δεδομένων και των παρεμβάσεων των συναδέλφων, οπότε μπορούμε να συνεχίσουμε τη διαδικασία. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, αυτό που προτείνω κύριε Σιγητά είναι να αρχίσουμε με μια προθεσμία για κατάθεση τροπολογιών όπως το είχαμε προβλέψει με τη διαδικασία για την έκθεσή σας και έπειτα στους συντονιστές θα μιλήσουμε και θα πούμε αν παράλληλα επιθυμούμε μέσα στο πνεύμα του άρθρου 91 του νέου μετά από την αλλαγή του κανονισμού αν επιθυμούμε να δεσμευτούμε στη διάρκεια της ψηφοφορία στην Ολομέλη για την έκθεσή σας για την εκπόνηση ενός ψηφίσματος. Τώρα θα ξεκινήσουμε, ε, μάλλον η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών θα πρέπει να, οι οποίε θα πρέπει να είναι μόνο ε, στα αγγλικά και ζητώ συγγνώμη εξ ονόματο των μη αγγλόφωνων ότι η προθεσμία λοιπόν είναι 28 Ιανουαρίου το, στις 12 το μεσημέρι. Θα τις εξετάσουμε στις 3 Φεβρουαρίου στη διάρκεια της έκτακτης μας συνεδρίασης και... Ε, τι συμβιβαστικές θα τις εξετάσουμε αν υπάρξουν στις 12 Φεβρουαρίου και θα τις ψηφίσουμε στις 13, ώστε αν είναι δυνατόν να περάσει από την Ολομέλεια στις 10 με 13 Μαρτίου, πράγμα που σημαίνει, αν κατάλαβα καλά, ότι θα είμαστε εντάξει και έτοιμοι πριν από την επόμενη τριμερή. καθώς το Συμβούλιο θα γίνει 20 με 23 Μαρτίου. Περνάμε τώρα στο σημείο 9, όπου θα εξετάσουμε τις τροπολογίες στην πρόταση κανονισμού του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού 718 του 1999 σε σχέση με μια πολιτική ρύθμιση της μεταφορικής ικανότητας των κοινοτικών στολών στην εσωτερική ναυσιπλοεία για την προώθηση των μεταφορών δια των πλωτών οδών. Εδώ πρόκειται για μια γνωμοδότηση που εμείς απευθύνουμε στην, στην Επιτροπή Μεταφορών, όπου εισηγείται είναι η κυρία Κόριν Βόρτμαν Κόλ. Η δική μας συντάκτρια γνωμοδότησης είναι η κυρία Γιούτα Στάινρουκ, στην οποία δίνω και το λόγο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όποιο εξέτασε τη γνωμοδότησή μου γνωρίζει ότι η πρότασή μου είναι σαφώς προς το συμφέρον των εργαζομένων Το Ταμείο βεβαίως ωφελεί και τις δύο πλευρές. Στα πλαίσια του εξυγχρονισμού των στόλων πρέπει ιδίω να ληφθεί υπόψη η κοινωνική και επαγγελματική κατάσταση των εργαζόμενων. ώστε και εργαζόμενοι αλλά και επιχειρήσεις να έχουν τη δυνατότητα τελικώς να μείνουν στη δουλειά, να μην μείνουν άνεργοι. και με πρόορες συνταξιδοτήσεις. Οι τεχνικές ρυθμίσεις επίσης παίζουν ένα ρόλο και το Ταμείο έχει και τον σκοπό να δώσει την ευκαιρία στα πληρώματα να λάβουν περαιτέρω κατάρτιση και για να υπάρχει και η δυνατότητα αυτή για περαιτέρω κατάρτιση είναι σημαντικό να χορηγούνται οι απαραίτητες πληροφορίες. Χαίρομαι για το γεγονός ότι και στις τροπολογίες της Ελίζαμπετ Σρόντερ και του κ. Ντεμπάκερ περιλαμβάνεται πάλι αυτή η ιδέα. Σημαντική προϋπόθεση τώρα για να δαπανηθούν τα χρήματα προς το συμφέρον και των εργαζόμενων αλλά και των επιχειρήσεων στον τομέα της ναυσιπλοείας είναι να δεσμευτούν και οι κοινωνικοί εταίροι για την ε, κατεύθυνση που θα λάβουν οι επενδύσεις γιατί αυτοί γνωρίζουν το επάγγελμα. Την επόμενη εβδομάδα θα συναντηθώ με τους κοιόδης συζήτητες για να συνεννοηθούμε. Όλες τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί τις δέχομαι και σε ό,τι αφορά την χορήγηση πληροφοριών αλλά και την προστασία του κλίματος που περιλαμβάνει ρητά στις τροπολογίες της κυρία Σρέντερ. Νομίζω ότι μπορούμε, θα μπορέσουμε ενδεχομένως να φτιάξουμε μια πρόταση που να την συνυποστηρίξουν όλοι. Ευχαριστώ. Α, τι ωραία λοιπόν. Ε, σήμερα άλλωστε είναι φεστιβάλ ντεμπάκερ από ό,τι βλέπω. Μα δεν είπα τίποτα, λέει ο κ. Ντεμπάκερ. Ναι, ναι, θα σα δώσω το λόγο αμέσω. Και μετά ο κύριο Ορή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ και την εισηγήτρια. Θα ήθελα να πω ότι ήδη, όπως έχω πει πάλι παλαιότερα, ότι η Κομισιόν έχει καταθέσει μια πολύ χρήσιμη πρόταση. Και το Ταμείο που πρόκειται να δημιουργηθεί θα βασίζεται και σε εξυγχρονισμό του στόλου, της εσωτερικής ναυσιπλοείας και σε μια ιδιαίτερη προσπάθεια τεχνικών προσαρμογών για την προστασία του κλίματος και ε, με σκοπό να επιταχυνθεί η προσπάθεια αυτή. Νομίζω ότι η κυρία Στάινρουκ θέλει ωστόσο να πάρει αυτό το ταμείο και να το κάνει κάπως κοινωνικό ταμείο, κάτι σαν κοινωνικό ταμείο, που δεν είναι σωστό το ταμείο είναι περιορισμένο και γι' αυτό πρέπει να φροντίσουμε ώστε οι δαπάνες να γίνονται με ιδιαίτερα προσεκτικό τρόπο. Με βασική κατεύθυνση τον εξυγχρονισμό του στόλου της εσωτερικής ναυσιπλοείας. Αυτό πρέπει να μας απασχολήσει πρωτίστως. Γι' αυτό και δεν με βρίσκουν σύμφωνο οι τροπολογίες 2, 3 και 6. Έχω καταθέσει εγώ ορισμένες τροπολογίες δικές μου, βασιζόμενος σε υφιστάμενα κείμενα, όπου κάνω μια προσπάθεια να επαναφέρω το κείμενο στην κατεύθυνση περισσότερο της προτάσεως της Κομισιόν. Διότι, όπως είπα, το Ταμείο πρέπει να εξυπηρετήσει κυρίως τον εξυγχρονισμό του στόλου της εσωτερικής ναυσιπλοείας. Ελπίζω ότι μεταξύ των σκιωδών εισηγητών θα μπορέσει να εξευρεθεί ένας κατάλληλος συμβασμός, γιατί είναι σημαντικό ο εσωτερικός τόλος να εξυγχρονιστεί και κάτι πρέπει να γίνει, γιατί ο σκοπός αυτός είναι πάρα πολύ σημαντικός. Ε, εσείς κύριε Ορή τώρα. Ευχαριστώ. Ο Ντέβιτ Κάσα είναι σκιώδης ηγητής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Ε, δυστυχώς είναι απασχολημένος σε άλλη συνεδρίαση αυτή τη στιγμή και γι' αυτό δεν μπορεί να είναι παρόν. Πολύ σύντομα λοιπόν έχω να πω τα εξή. Ο συναδελφός μου δέχεται την αρχική πρόθεση της Κομισιόν να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής στο άρθρο 8 και τονίζει επίσης ότι βοθήσεις της κρίσεως αλλά και της πάνιδας των πόρων ο τομέας που έχει διέλθει μέσα από πολύ δυσχερείς περιστάσεις έχει ανάγκη να υποστηριχθεί. Και γι' αυτό ο συναδελφός υποστηρίζει την πρόταση της Κομισιόν. Όμως εκφράζει ορισμένες επιφυλάξεις όσον αφορά τις προτάσεις της ηγήτριας όπου φοβείται ότι ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις από τις προτάσεις της εισηγήτριας. Και γι' αυτό έχει καταθέσει ο ίδιος ορισμένες τροπολογίες και αφετέρου δεν υποστηρίζει όλες τις τροπολογίες της Όμως, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα δεν έχει συζητήσει ακόμα με λεπτομέρεια το θέμα. Πρόκειται λοιπόν για ένα πρώτο προβληματισμό του συναδέλφου μου David Κάσα. Ε, αυτό είναι το νόημα των λόγων που σας είπα. Η πρόεδρος, κυρία Μπερές. Άλλος κανείς ή άλλη καμία. Όχι, η Κομισιόν. Μάλιστα. Εσείς. Ο κύριος Θεολογίτης. Μάλλον όμως μου φαίνεται προέρχεστε από χώρα που έχει σχέση με την ε, εξωτερική ναυσιπλοεία. Γιατί η ναυσιπλοεία είναι στη θάλασσα και όχι στην εσωτερική. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Γνωρίζετε ότι η μόνη εσωτερική ναυσιπλοεία που μπορώ να θυμηθώ σε σχέση με την Ελλάδα είναι αυτή στον ε, ποταμό Αχέροντα, όπου ο χάρος περνάει τις ψυχές ε, απέναντι στον κάτω κόσμο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντως χαίρεται για την ταχεία απάντηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την πρότασή της, που έχει στόχο να διευκολύνει την χρήση του Ταμείου που έχει δημιουργηθεί από τον ίδιο τον κλάδο, από τους ε, πλειοκτήτες μικρών και μεσαίων σκαφών, όταν χρειάστηκε να μειώσουμε την χωρητικότητα. Ελπίσαμε λοιπόν να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί και τώρα σε παραπάνω από 10 χρόνια που έχει δημιουργηθεί το ταμείο αυτό αποδείχθηκε ότι είναι δύσκολο να χρησιμοποιηθεί. Και για το λόγο αυτό πρόθεσή μας είναι να διευκολύνουμε την χρήση του ταμείου, όπως άλλωστε το εξήγησε και η συγκήτρια, σε περίοδους κρίσεως όπως τώρα και βέβαια σε χρόνους κάποιων αλλαγών, αναγκών προστασίας του κλίματος, μειώσεως των ε, εκπομπών αλλά και τεχνολογικών αλλαγών. Αυτή είναι η βασική στόχη της προτάσεως της Κομισιόν. Εμείς βλέπουμε πάντως ότι οι περισσότερες τροπολογίες δέχονται την κατεύθυνση αυτή και την υποστηρίζουν. Τι δεχόμαστε λοιπόν. Έχουμε όμω ορισμένε επιφυλάξει όσον αφορά μια διαγραφόμενη τάση να πάει να γίνει κοινωνικό ταμείο. Δεν είναι όμω αυτός ο σκοπός του ταμείου. Κοινωνικό ταμείο θα ήταν πολύ ωραίο και καλοδεχόμενο, χρειάζεται όμω διαφορετική οργάνωση, την οποία δεν διαθέτει το συγκεκριμένο εργαλείο, στο οποίο έχουν συμβάλει, όπως είπα, οι φορείς του κλάδου, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε εμεί είναι να εξασφαλίσουμε ότι θα χρησιμοποιηθεί από τον κλάδο σύμφωνα με τι ανάγκε του και να το ανοίξουμε. Αυτά λοιπόν παρακαλώ λάβετε υπόψη σας και ας μην κινηθούμε προς μια κατεύθυνση που δεν θα διευκολύνει, αλλά μάλλον θα παρεμποδίσει την χρήση του Ταμείου. Αυτό είναι το μοναδικό σχόλιο που επιθυμώ να κάνω. Και επαναλαμβάνω τι ευχαριστίε μου προ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι έχουμε την ελπίδα ότι σε συνεργασία με την Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου θα μπορέσουμε να επιτύχουμε συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση ήδη μέσα στην τρέχουσα κοινοβουλευτική θητεία εποφελία του κλάδου. Ευχαριστώ. Κανείς άλλος. Παρακαλώ κυρία Συγκήτρια. Υπενθυμίζω ότι η ίδρυση του Ταμείου είχε την πρόθεση να φτιάξει ένα κοινωνικό ταμείο που όμως λόγω διαφόρων συνθήκων πλαισίων δεν χρησιμοποιήθηκε τελικά. Εμείς εδώ είμαστε Επιτροπή Απασχολήσεως που υποτίθεται ότι παρακολουθούμε την εφαρμογή των συνθήκων πλαισίων έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον αυτό το ταμείο και εφόσον έχουμε και σε άλλους οικονομικούς κλάδους ε, αναδιαθρώσεις και μιλούμε για αναδιαθρώσεις, για εξυγχρονισμό για μείωση ενδεχομένως των στόλων. Εμείς ως Επιτροπή Απασχολήσεως οφείλουμε όντως να λάβουμε υπόψη την κατάσταση των εργαζομένων. Είναι απαραίτητη λοιπόν η κατάρτιση, η απόκτηση δεξιοτήτων ε, όταν μιλούμε για μείωση των στόλων, επίσης η μετάβαση στην συνταξιδοτική ηλικία, χορήγηση ε, πληροφοριών, συμβουλών, μετεκπαίδευση είναι ενδιαφέρον ότι και η Επιτροπή Περιβάλλοντος, περιβάλλον το λέτε εσείς ως στόχο, έτσι το αναφέρετε ως στόχο, δεν θεώρησε απαραίτητο να, να συντάξει γνωμοδότηση γιατί βλέπει, εκεί, γιατί βλέπει και η ίδια αυτή η Επιτροπή ότι εδώ ο κύριος στόχος είναι τα κοινωνικά. Αυτές θεωρώ ότι είναι οι προθέσεις λοιπόν και ως Επιτροπή Απασχολήσεως επαναλαμβάνω θεωρώ ότι είναι καθήκον μας τις προτάσεις αυτού του είδους της Κομισιόν να τις ελέγχουμε και από την άποψη της καταστάσεως των εργαζομένων και των επιπτώσεων στους εργαζομένους. Και αυτοί που ξεκίνησαν το Ταμείο μου δήλωσαν σαφώς ότι αρχικά και αρχήθεν δηλαδή πρόθεσή τους ήταν να είναι και κοινωνικό ταμείο. Μάλιστα λέει η πρόεδρος. Επί της βάσης αυτής θα εξετάσουμε τις τροπολογίες συμβιβασμού στις 12 Φεβρουαρίου. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις 13 και η Επιτροπή Μεταφορών θα ψηφίσει στις 20 Φεβρουαρίου στη βάση του άρθρου 50. Ολοκληρώσαμε τη συζήτηση αυτού του θέματος και ερχόμαστε τώρα στο υπαριθμό 10. Το σημείο 10 αφορά την πρόταση κανονισμού, έκθεση για την οποία κατ' ουσίας αρμόδια είναι η Επιτροπή ΕΚΟΝ, με θέμα τις στατιστικές σχετικά με τη διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών. Έχουν κατατεθεί 18 τροπολογίες και θα σας τις παρουσιάσω για να τις εξετάσουμε. Μάλιστα 8 από τις 10 τις κατέθεσα εγώ. Σε ό,τι αφορά την τροπολογία 10 της κυρίας Κορνέλησεν δεν έχω πρόβλημα, ούτε και με την τροπολογία 10, γιατί εμπλουτίζουν ε, το κείμενο με πολύ καλό τρόπο. Τροπολογία 11 του κυρίου Τσάμπα Όρη. Φοβάμαι ότι τροποποιεί το στόχο του κειμένου γιατί τροποποιεί την ανάγκη στατιστικών που είναι απαραίτητες για τα θέματα της οικονομικής ε, δραστηριότητας. Θα μετατρέπει σε θέμα κοινωνικής πολιτικής, κάτι που είναι διαφορετικό. Θα ήθελα λοιπόν ο κύριος Όρη να μου εξηγήσει την τροπολογία 12 επίσης, γιατί φοβάμαι ότι η τροπολογία αυτή περιορίζει κάπως τις φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν συμφωνώ με αυτό. Δεν έχω πρόβλημα με την τροπολογία 13 της κυρίας Κορνέλισεν που θέλει να ενισχύσει τη συμβολή αυτών των ε, στατιστικών στην οικονομική διακυβέρνηση. Η τροπολογία 14 λέει ότι τα κράτη-μέλη δεν θα πρέπει να διαβιβάζουν αλλά να κοινοποιούν τα κατάλληλα στοιχεία. Διαρωτώ με πως έτσι αποδυναμώνουμε την υποχρέωση των κρατών μελών. Κάτι που δεν με βρίσκει φωνή Με την τροπολογία 15 δεν έχω πρόβλημα. Ούτε και με την τροπολογία 16 του κύριου Κρόιτσμαν. Αντίθετα, θα πρέπει να γίνει μια επιλογή μεταξύ των τροπολογιών 17 Κρότσμαν και 18 Ορί. Νομίζω ότι η τροπολογία 18 του κυρίου Ορί είναι πιο ακριβής, γιατί μιλάει για την διαβίβαση των στατιστικών στις αρμόδιες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στην Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής. Είναι πιο ακριβής αυτή η τροπολογία και θα παρότρινα ένα από του δύο συγκεκριτές να αποσύρει τη δική του. Τροπολογία 19. Ο κύριο Κρόισμαν θέλει να δώσει την ευκαιρία στα κράτη-μέλη να δώσουν εξηγήσει ε, για την κατάσταση. Νομίζω ότι παρά είναι γενναιόδωρο και επίκη ο κύριο Όρη σε σχέση με του ε, στόχου που επιδιώκουμε. Η τροπολογία 20 και 21 είναι παρόμοιε και δεν με βρίσκουν σύμφωνοι. Σε ό,τι αφορά την τροπολογία 22 του Τσαμπόρη δεν έχω πρόβλημα. Θα ήθελα όμως να μου εξηγήσει τι εννοεί με την τροπολογία 23 ο κύριος Σόρη. Για να είμαστε σίγουροι ότι ευθυγραμμίζεται με τους στόχους μας. Η τροπολογία 24 του κυρίου Κρόιτσμαν είναι πιο γενναιόδορη προς τα κράτη-μέλη και περιορίζει τη δυνατότητα παρεμβάσεων με την επιβολή προστήμων. Δεν συμφωνώ. Αντίθετα, η τροπολογία 25 ε, του κυρίου Κρόιτσμαν επαναφέρει μία παλιά μας ιδέα που λέει ότι τα έσοδα από τα πρόστιμα προορίζονται για μέτρα προστόνωση των επιπέδων απασχόλησης και εκπαίδευσης, ειδικά μεταξύ των νέων. Πολύ εύστοχη τροπολογία και θα την υποστηρίξω. Επίσης, τροπολογία 26 της κυρίας Κορνέλισον προσδιορίζει τις εθνικές αρχές μεταξύ άλλων που μπορούν να ενεργοποιηθούν στα πλαίσια του κανονισμού και επίσης ε, συμφωνώ με την έκθεση της κυρίας Κορνέλισε. 18 λοιπόν συνολικά τροπολογίες, ολόκληρος κατάλογος ε, με τροπολογίες και τώρα θα ακούσουμε τους συντάκτες. Πρώτα κυρία, ο κύριος ε, Τσάμπα Όρη. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, ε, με τις τροπολογίες Προσπάθησα να βελτιώσω την ε, έκθεση. Όσον αφορά την παράγραφο 3, προσπαθώ να κάνω μία σύντομη προσθήκη. Εδώ γίνεται μία παρήθμιση για τις περιπτώσεις όπου η Κομισιόν μπορεί να κάνει επαλήθευση. Αυτό είναι καλό. Προσθέτω πως ε, η Κομισιόν θα πρέπει να κάνει την ανάλυση αυτή με, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Γι' αυτό γιατί ήθελα απλά να διευκρινίσω πως οι δυνατότητες παρέμβασης της Κομισιόν δεν μπορούν να είναι απεριόριστες. Θα πρέπει να περιορίζονται Πώς είπατε, για ποια παράγραφο μιλάτε, την 23, μα δεν υπάρχει. Μιλάτε για την τροπολογία 23. Ναι, τροπολογία 23, ναι, έκανα λάθος. Ήθελα να πω τροπολογία και είπα παράγραφο. Δεν ήταν η παράγραφος 23, ήταν η τροπολογία 23. Εγώ δεν έχω πρόβλημα για την 23. Εγώ πιστεύω πως η Κομισιόν μπορεί να κάνει όλες τις ε, σχετικές έρευνες. Δεν θέλω να μειώσω την αρμοδιότητα της Επιτροπής, αλλά να οριοθετήσω τις αρμοδιότητές της. L'amendement 11 euh,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 η ουσία δεν είναι διαφορετική. Αλλά δεν είναι και κεντρικό θέμα. Δεν θα τσακωθούμε γι' αυτό. Πιστεύω πως κατ' ουσίαν δεν υπάρχουν δυσκολίες για το κείμενο. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες ε, διαφορές διατύπωσης. Ήθελα απλά να διατυπώσω πιο συγκεκριμένα ε, να συζητήσουμε αυτές τις τροπολογίες με εσάς που τις υποβάλλατε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εκ μέρους του κυρίου Κρότσμαν, λέει κυρία Χίρς, να σας πω λίγα λόγια για το πώς βλέπει τις τροπολογίες ο ίδιος. Και πρώτα επιθυμεί βέβαια να ευχαριστήσει για την συνεργασία καθώς επίσης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υποβολή της προτάσεως. Αναμένει ταχεία συμφωνία με το Συμβούλιο. Βρίσκει ότι είναι πολύ σημαντικές οι ορθές στατιστικές και είναι πολύ βαριές οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις όχι μόνο η Ελλάδα αλλά και άλλες χώρες και η Γερμανία στο παρελθόν έχουν υποβάλει, έχουν τέλος πάντων ε, τροποποιήσει τις στατιστικές προς όφελός τους. Η Κομισιόν έχει περιλάβει και ρυθμίσεις για να επιτρέπει τους εμμυρογνώμονες να εξετάζουν τα στατιστικά δεδομένα επί τόπου, όμως αυτό το έχει απορρίψει το Συμβούλιο. Τώρα σε περιπτώσεις ελλείψεων μπορούν να γίνονται έλεγχοι επιτόπου σε χώρες μέλη. Δεχόμαστε την διεύρυνση του πεδίου εφαρμογή λόγω της ανάγκης αποκατάστασης μακροοικονομικών ισορροπιών, διότι δεν μπορεί να υπάρξει πρόοδος χωρίς σύγκριση των οικονομιών και αυτή θα λειτουργήσει μόνο στη βάση πλήρων και αξιόπιστων στατιστικών δεδομένων. Λίγα λόγια ακόμα για το βαθμολόγιο, scoreboard, όπου απορρίπτουμε την επιβάρυνσή του με κοινωνικούς δείκτες, που δεν είναι απαραίτητη για την μακροοικονομική σταθερότητα. Ούτως ή άλλως η Κομισιόν σε περίπτωση σοβαρών ανισορροπιών κάνει ειδικέ μελέτε. Θέλουμε λοιπόν ένα ξεχωριστό μη δεσμευτικό βαθμολόγιο. Ο κ. Κρότσμαν βλέπει ανάγκη να διευκρινιστεί επίσης το άρθρο 9 παράγραφο 5 όπου σε περιπτώσεις προστήμων η Κομισιόν θέλει να μπορεί να, τις, να συμπράττει τις ποινές αυτές η ίδια. Η Κομισιόν θα πρέπει όμως να εξηγήσει ποια είναι η νομική τη βάση, ζητεί ο κ. Κρότσμαν και ο οποίος υποστηρίζει την πρόταση της Κομισιόν οι χρηματικές ποινές να εφαρμόζονται σε όλες τις χώρες μέλη και τα ποσά αυτά να καταλήγουν στον ενωσιακό προϋπολογισμό. Δεν βλέπει κανένα λόγο να γίνει οποιαδήποτε διάκριση μεταξύ χωρών ευρώ, ζώνης ευρώ δηλαδή, και άλλων χωρών εκτός. Ε, Θέλει άλλος καλύτερο λόγο. Όχι. Οπότε να δώσω το λόγο στον Άλε Καπέκα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε καθυστερήσει κάπως, γι' αυτό σας θέλω παρακαλώ να είστε σαφής και λακωνικός. Ευχαριστώ. Ο κανονισμός αυτός είναι απαραίτητος για να εξασφαλιστεί η ποιότητα των στατιστικών στη διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών, όπως είπαν και οι προλαλήσαντες. Χαιρετίζουμε λοιπόν τις ε, τροπολογίες γιατί δεν αλλάζουν την ουσία του κανονισμού, αλλά αντίθετα ενισχύουν κάποια στοιχεία του. Και ιδιαίτερα το πλαίσιο ε, α, της ποιότητας των στατιστικών. Έχω κάποια σχόλια που αφορούν περισσότερο την διατύπωση, την ακρίβεια της διατύπωσης και όχι τόσο την ουσία. Για παράδειγμα, η τροπολογία 14 που προσπαθεί να αντικαταστήσει το transmitting of data, τη διαβίβαση των ε, ε, δεδομένων στην Επιτροπή από τον όρο communicating, να κοινοποιήσει. Ε, εμείς προτιμούμε τον όρο transmitting, διαβίβαση από τα κράτη-μέλη στην Επιτροπή. Είναι πιο δόκιμος ο, ρόλος αυτό, ο όρος αυτός, τον transmitting από το communicating. Άρα είναι θέμα τεχνικό ίσονο Σε ό,τι αφορά τα πρόστιμα, μετά από σκέψεις και ανάλυση, περιλάβαμε στον κανονισμό την ε, δυνατότητα επιβολής κυρώσεων. Στα κράτη-μέλη που έσκεμμένα ή λόγω ε, αμέλειας ε, σοβαρής δεν χορηγούν ποιοτικά στατιστικά στοιχεία. Βάζουμε τις κυρώσεις ως αποτρεπτικό στοιχείο για να αποτρέψουμε τα κρατημέλη από τον υποβάλλον ασφαλμένα στατιστικά. Δεν ξέρω πώς θα χρησιμοποιηθεί στην πράξη τελικά αυτό το άρθρο για την επιβολή κυρώσεων ή προστήμων, αλλά θα θέλαμε να παραμείνει στον συντονισμό, άλλωστε συνάδει με κανονισμούς αντίστοιχους σε άλλους τομείς. Άλλωστε δεν υπερβαίνουν το 0,05% του ΕΑΕΠ του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους. Επίσης θα θέλαμε να προσδιορίσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια τους κανόνες για τα πρόστιμα και το ύψος τους. Γιατί Υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα ε, κακής υποβολής στατιστικών ή ε, εύρους ε, αμέλειας. Θα πρέπει να θεσπίσουμε κριτήρια λοιπόν για τον προσδιορισμό του ποσού των προστήμων που αναφέρονται στο άρθρο. Αυτά. Ευχαριστώ. Τέθηκε και μία ερώτηση για το κατά πόσο θα πρέπει να θεσπιστεί δικός κανονισμός για την Ευρωζώνη. Ο κανονισμός αυτός ισχύει για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχουμε προβλέψει ξεχωριστό κανονισμό ή ξεχωριστά πρόστιμα για τις χώρες Ευρωζώνης. Το άρθρο αυτό θα πρέπει να ισχύει για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μάλιστα σχετίζεται με την τροπολογία 5 Δεν καταλαβαίνω γιατί τα έσοδα από τα πρόστιμα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν μόνο για τις χώρες της Ευρωζώνης ή μόνο στις χώρες της Ευρωζώνης. Θεωρούμε ότι ο κανονισμός ισχύει για όλα τα κράτη-μέλη. Θέλουμε να κάνουμε διακρίση μεταξύ χώρες εντός και εκτός Ευρωζώνης. γιατί προβλήματα και στις χώρες εκτός Ευρωζώνης μπορούν να επηρεάσουν όλες τις υπόλοιπες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θέλουμε λοιπόν να περιορίσουμε το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού μόνο στις χώρες της Ευρωζώνης ή να περιορίσουμε το πεδίο εφαρμογής συγκεκριμένου άρθρου μόνο στις χώρες της Ευρωζώνης. Πολύ ωραία. Θα λάβουμε υπόψη τις παρατηρήσεις σας. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτές. Θα τις λάβουμε υπόψη και θα συντάξουμε ενδεχόμενες ε, συμβιβαστικές τροπολογίες έτσι ώστε να συνδεθούν οι αρχικές μου προτάσεις με αυτές των συντακτών των τροπολογιών, ιδιαίτερα για το τελευταίο σημείο που αναφέρθηκε. Νομίζω ότι με τους συντάκτες των τροπολογιών θα μπορέσουμε να εξετάσουμε εκ του σύνεγγυς της τροπολογίες όπως θα πρέπει και να δούμε μάλλον αν θα πρέπει να μπουν ή όχι στο τελικό κείμενο διατηρώντας ε, το πνεύμα της πρότασης της Κομισιόν και την βούληση να συμβάλλουμε έτσι στην ενίσχυση της διαδικασίας όσον αφορά τις μακροοικονομικές ανισορροπίες. Θα εξετάσουμε λοιπόν τις συμβιβαστικέ αυτές στη συνεδρίασή μας, στην έκτακτη αυτή συνεδρίαση της 3ης ε, Φεβρουαρίου και θα ε, ψηφίσουμε την ίδια συνεδρίαση γιατί η ΕΚΟΝΑ ε, θα ψηφίσει τον Απρίλιο γι' αυτό. Ε, πάντοτε ε, βλέπουμε, συνεχίζουμε να έχουμε καθυστερήσει σε σχέση με την ημερήσια μετέταξη, να χαιρετήσω τους υπεύθυνους των διαφόρων οργανισμών και κέντρων. Ωστόσο θα δώσω γρήγορα το λόγο στην Νατάλια Γιαζοβιέσκα, για να μας ε, αναφέρει τις εξελίξεις ε, στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο με θέμα την επιβολή της οδηγίας 9671 για την απόσπαση των εργαζομένων. Θα έχετε καταλάβει δυστυχώς κύριε Συγκήτρια ότι θα πρέπει να είστε πολύ λακωνικοί για να μας δώσετε τις πληροφορίες για αυτό το πρώτο τριμέρι διάλογο. Έχω ερώτηση. Να είμαι άκρος τηλεγραφική ή απλώς τηλεγραφική. Okay, θα προσπαθήσω. Είχαμε τον πρώτο τρίλογο για την οδηγία που αφορά την απόσπαση των εργαζομένων. Δυστυχώς ε, δεν έχουμε ακόμη εντολή για τη διαπραγμάτευση, οπότε είναι όλο πρόκαταρκτικές αυτές οι συμφωνίες. Μιλήσαμε για το άρθρο 1, παιδιοφαρμογής, άρθρο 2, ορισμοί, άρθρο 4, ο ε, ε, ρόλος Ινστιτούτων και Γραφείων Σύνδεσης και άρθρο 5 πρόσβαση στις πληροφορίες. Σε ό,τι αφορά το πρώτο άρθρο είχαμε καλές και επικοδομητικές συζητήσεις. Καταλήξαμε σε κοινέ ε, θέσεις για 90% της διατύπωσης αλλά δεν είχαμε χρόνο για να ασχοληθούμε με ένα από τα τελευταία εδάφια του άρθρου 5. Άρθρο 1 λοιπόν. Πεδίο εφαρμογή οδηγία. Καταλήξαμε συμβαστικό κείμενο με βάση τι τροπολογίε του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου. Δεν έγιναν αλλαγέ στο πεδίο εφαρμογή οδηγία. Ε, αναφέρεται ότι η οδηγία εφαρμογή δεν τροποποιεί την αρχική οδηγία του 1996. Σε ό,τι αφορά ε, τη, την οδηγία αυτή, α, ε, αναφέραμε ότι τηρεί το διεθνέ δίκαιο. Επίσης, τηρούνται οι υποχρεώσεις που απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις που έχουν υπογραφεί. Σε ό,τι αφορά το άρθρο 2 για τους ορισμούς, ε, είχαμε την, ε, το ορισμό για το ιδιαίτερο Ινστιτούτο, για τις ε, συγκεκριμένες αρμοδιότητες κάποιων ιστιτών. Σε ό,τι αφορά ευθυγράμμιση των οργάνων συνεργασίας που αναφέρονται στο έκτο τμήμα της οδηγίας για, την για τη διασυνοριακό χαρακτήρα κυρώσεων και προστήμων. Επίσης ε, για τη... τα γραφεία σύνδεσης και τα διάμεσα Ινστιτούτα είχαμε είχαμε συμβαστικές λύσεις. Η αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμπληρώθηκε με την υποχρέωση των κρατών μελών να εξασφαλίσουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων και αναφέρεται ότι τα γραφεία σύνδεσης ε, μπορούν να δίνουν πληροφορίες για τους όρους ε, πρόσληψης στα κράτη-μέλη. Το Συμβούλιο εξαιτία σημαντικών διοικητικών διατυπώσεων δεν συμφώνησε να δοθεί αρμοδιότητα και παρακολούθηση στα γραφεία σύνδεσης ε, για το κατά πόσο τηρούνται οι αρχές πρόληψης. Άρθρο 5. Πρόσβαση στην ενημέρωση. Και εδώ καταλήξαμε σε συμβαστική λύση για το πρώτο τμήμα του άρθρου 5. Το Συμβούλιο συμφώνησε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για, ώστε οι όροι πρόσληψης να δημοσιεύονται σε μια ενιαία ιστοσελίδα. Επίσης, Είχαμε αναφορά του κειμένου τη οδηγία για την ελεύθερη διακίνηση των εργαζομένων και σχετική έκθεση της Edith Bauer. Θα πρέπει οι πληροφορίες να γίνονται στη γλώσσα της χώρας υποδοχής ε, και φυσικά να ληφθεί υπόψη η υπηκότητα των ε, εργαζομένων. Το Συμβούλιο συμφωνεί τα κράτη-μέλη να δημοσιεύσουν πληροφορίες και για τι διαδικασίε ε, υποβολή κυρώσεων σε ανέντιμου εργοδότες. Βέβαια θα συνεχιστούν οι διαβουλεύσεις στο Συμβούλιο. Άλλαξε κάπως η παράγραφος για την ευθύνη των κοινωνικών εταίρων για τη δημοσίευση ε, πληροφοριών για τις συνθήκες ε, πρόσληψης. Το κείμενο συμβασμού λέει ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι πληροφορίες για τις ε, συνθήκες πρόσληψης των κοινωνικών εταίρων θα πρέπει να είναι δημοσίως προσιτές και γι' αυτό θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά και η κοινωνική Ε, Θα έχουμε την επόμενη, τον επόμενο διάλογο ε, στις 23 ε, Ιανουαρίου για τα θέματα και των εφαρμοστικών ε, διατάξεων. Ναι, όντως, αύριο θα είναι ο τριμερής διάλογος για το άρθρο 3, οπότε αύριο θα αρχίσει η σοβαρή συζήτηση. Υπάρχουν, Υπάρχουν ερωτήσεις, κατανόησεις ή παρατηρήσεις. Όχι. Ωραία, λοιπόν, στην επόμενη μας συνεδρίαση θα μας ενημερώσετε για την αυριανό τριμερή διάλογο. Ολοκληρώθηκε λοιπόν και αυτό το σημείο της ημερής διάταξης. Ευχαριστώ πολύ τους τέσσερις ε, διευθυντές των οργανισμών που περίμεναν υπομονετικά, αλλά έγκυκε η ώρα να προχωρήσετε στην παρουσίαση των προγραμμάτων εργασιών σας για το έτος 2014. Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχηθώ καλή χρονιά εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και με αυτή την ευκαιρία θα πρέπει ε, να σας πω ότι χαίρομαι που μπορούμε να ανταλλάξουμε απόψεις για τα έγγραφα τα οποία έχουν ήδη δοθεί στα μέλη της Επιτροπής. Σας προτείνω λοιπόν να ξεκινήσουμε με την κυρία Κρίστα Τζέντλετ Στίκ, που είναι διευθύντρια του Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία. Έχετε το λόγο. Thank you very much, uh, Madam Chair, and also wish you all... Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Σας εύχομαι υγιές και επιτυχές έτος, ένα πολύ σημαντικό έτος για την Ευρώπη. Στα έγγραφα που έχετε λάβει τονίζονται κάποιοι τομείς προτεραιότητας ξεκινώντας από την εργασία μας για την ε, online ε, εκτίμηση κινδύνου, αξιολόγηση κινδύνου. Θα το έχετε ήδη ακούσει οι περισσότεροι. Είναι αυτό το γενικό εργαλείο για τις μικρές ε, μετακινούμενες εταιρείες που έχουμε αναπτύξει και τώρα θέλουμε να επιτύχουμε να κινητοποιήσουμε περαιτέρω εξελίξεις σε επίπεδο κράτους μέλους και τομέα και είμαστε ήδη στην πολύ καλή κατάσταση όπου 12 τέτοια εργαλεία ε, για την αξιολόγηση κινδύνου είναι ήδη βρίσκονται ε, ανακοινωμένα επιγραμμικά ε, και αυτό απευθύνεται στις μικρές και στις μικροεπιχειρήσεις. Όπως γνωρίζετε έχουμε λάβει από πλευρά των οργανισμών όλα αυτά τα εργαλεία να γίνονται σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και στην ανάπτυξή τους και προβλέπουμε του χρόνου ε, ακόμα 60 εργαλεία αξιολόγησης κινδύνου σε διάφορες χώρες και τομείς. Δεύτερον, θα ήθελα να στραφώ σε ένα, μία από τις ναυαρχίδες μας στον τομέα της ε, συνειδητοποίησης. Έχουμε διεξάγει την εκστρατεία του 2012 με 2013 και με το σύνθημα «Συνεργαζόμενοι για την πρόληψη του κινδύνου» και συνεργασία για την πρόληψη του κινδύνου και μπορέσαμε να κάνουμε μια πολύ καλή και θετική εταιρική σχέση. Αυτή η διετής εκστρατεία διαρκώς ε, μεγαλώνει, διευρύνεται. Έχουμε τώρα 87 επίσημους εταίρους της εκστρατείας αυτής και το 2014 και 2015 θα συνεχίσουμε με μια νέα διετή εκστρατεία, γιατί πρόκειται για ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει όλα τα κρατημέλη, όλες τις εταιρείες. Το σύνθημα είναι υγιής χώρος εργασίας, διαχείριση του στρες. και το feedback από τα εταίρους μας στα κατημέλη είναι πολύ θετικό. Η ανταπόκριση δηλαδή είναι πολύ θετική και προσβλέπουν στη συμμετοχή, στην αύξηση της συνειδητοποίησης. Ε, το θέμα αυτό είναι ζήτημα για τις εταιρείε και πάλι θέλουμε να στηρίξουμε τα κρατημέλη με το πακέτο της εκστατείας μας όπου ε, θα στηρίξει τη διοργάνωση εκδηλώσεων στα κρατημέλη. Αυτό λοιπόν για το 2014 με 16 όπου εργαζόμαστε για το θέμα των ψυχοκοινωνικών κινδύνων. Δεύτερον, θα ήθελα να επανέλθω σε ένα project που ξεκινήσαμε, ένα πιλωτικό πρόγραμμα για το Ευρωκοινοβούλιο ε, για την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας στο πλαίσιο ενός ε, γυράσκοντος εργατικού δυναμικού. Ευχαριστούμε την ε, κυρία Μπερές γιατί κάναμε μια ημερίδα της μισής μέρας και παρουσιάσαμε εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο τα πρώτα μας πορίσματα καθώς και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε μέχρι το 2015 διότι ο στόχος μας είναι να είμαστε σε θέση να προβούμε σε συστάσεις επί τη βάση της εργασίας μας στη διάρκεια αυτών των δύο ετών. Συστάσεις για το τι υπάρχει για να μπορέσει κανείς να διαχειριστεί το γυράσκον εργατικό δυναμικό που υπάρχουν ανάγκες σε επίπεδο κρατών μελών αλλά βέβαια σε τομεακό επίπεδο και στο επίπεδο της επιχείρησης. Το επόμενο θέμα είναι η δημοσίευση μιας σύντομης έκθεσης για την μείωση των κινδύνων στον τομέα υγείας και ασφάλειας για τις ε, γυναίκες στην ε, εργασία. Πρόκειται για μια σημαντική δημοσίευση επί της οποίας εργαζόμαστε εδώ και πάνω από 1,5 χρόνο και φυσικά θα προσφέρει συγκεκριμένες πληροφορίες για τα θέματα της υγείας των γυναικών και τον αντίκτυπο της εργασίας στην υγεία των γυναικών. Και ε, βέβαια ε, και κάτι αντίστοιχο ε, και για τους άντρες θα γίνει αργότερα. Τώρα, στρατηγικό σχεδιασμό των εργασιών του οργανισμού. Έχουμε συντάξει στρατηγικό πρόγραμμα εργασιών 2014 με 2020 Έχουμε αναπτύξει ένα πολυετές στρατηγικό πρόγραμμα τα τελευταία δύο χρόνια. Ε, δεν έχει υπάρξει και τόση συζήτηση τελικά, αλλά θα εργαστούμε επί πέντε βασικών τομέων, προβλέποντας τις αλλαγές και τους νέους αναδυόμενους κινδύνους, ε, εργαλεία για τη διαχείριση, την αύξηση της γνώσης, της συνειδητοποίησης, και αντιμετώπιση των προκλήσεων και φυσικά σε όλους αυτούς τους τομείς θα χρησιμοποιήσουμε τη δικτύωσή μας αλλά και την επικοινωνία με τις εταιρείες ώστε να μπορέσουμε να διαδώσουμε όσο γίνεται περισσότερο το μήνυμα για το πόσο σημαντικό είναι να έχουμε ασφάλεια και υγεία στο χώρο εργασίας σας στην Ευρώπη. Τώρα έρχομαι περισσότερο στον οδικό χάρτη, την εφαρμογή αυτού για να σας πω ότι στις 20 Δεκεμβρίου 2013 το το Συμβούλιο των Υπουργών έκανε μια συμφωνία ανάμεσα στην Ισπανία και στον οργανισμό μας, δηλαδή θα πάω στην Μαδρίτη σε λίγες μέρες για να υπογράψουμε τη συμφωνία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να έχουμε ένα ε, ρυθμισμένο πλαίσιο για τον οργανισμό μας, αλλά και πάλι σε σχέση με τον οδικό χάρτη και τη διαχείριση του προπολογισμού του οργανισμού μας, ε, μετακινηθήκαμε σε ένα νέο ε, κτίριο στον Μπιλμπάο και με βάση δύο κριτήρια όταν ε, ξεκινήσαμε αυτό το εγχείρημα. Το πρώτο να εξοικονομήσουμε χρήματα και δεύτερον να βελτιώσουμε τις συνθήκες εργασίας. Τα καταφέραμε και τα δύο. Βέβαια δεν είναι κατάλληλη στιγμή για την αγορά, οπότε εξοικονομούμε 40% από το ενίκιο που πληρώνουμε και έχουμε ταυτόχρονα πολύ περισσότερο χώρο για το προσωπικό μας καθώς και τη δυνατότητα να διοργανώνουμε συνεδριάσεις με τους φορείς μας και πάλι δηλαδή εξοικονομούμε χρόνο και χρήμα. Αυτή είναι η αναφορά μου και σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ και για αυτή την αίσθηση χρονισμού που έχετε, που ήταν τελεία, διότι μιλήσατε ακριβώς όσο έπρεπε. Και τώρα θα δώσω το λόγο για πρώτη φορά στον Ιωακίμ Τζέιμς Και Σας περιμέναμε πολύ καιρό κατά κάποιο τρόπο και τώρα πολύ χαιρόμαστε που σας έχουμε εδώ ως ενεργό πλέον διευθυντή αυτού του κέντρου για την ανάπτυξη της επαγγελματική κατάρτισης. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και πρώτα θα ήθελα να ανταποδώσω τις ευχές για το 2014 και σε εσά και στα μέλη σας. Είμαι στην 97η μέρα μου στο Σεντεφόπ και στο τέλος της εβδομάδας θα έχω συμπληρώσει 100 μέρες και ελπίζω ε, η αξιολόγηση που θα μου γίνει να είναι θετική. Στη Θεσσαλονίκη λοιπόν βρήκα έναν οργανισμό πραγματικά πάλλοντα που νομίζω ότι παίζει όλο και μεγαλύτερο ρόλο για την αντιμετώπιση των υψηλών ποσοστών ανεργίας, ιδίως των νέων. Η βελτίωση λοιπόν της δυνατότητας απασχόλησης των νέων ε, δίνει ιδιαίτερο στόχο στην μεταρρύθμιση των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης στο λεγόμενο empowering των ε, πολιτών για να υπάρξει μεγαλύτερη απασχόληση. Στα τέλη του περασμένου έτους οι εξωτερικοί αξιολογητές για το έργο του ΣΕΝΤΕΦΟΠ που καλύπτεται έτη από 2007 έως 2012 επιβεβαίωσαν την πρώτη μου θετική εντύπωση του οργανισμού διότι είπαν ότι το ΣΕΝΤΕΦΟΠ υπήρξε πολύ επιτυχημένο στην εφαρμογή των στόχων του, στην επίτευξη των στόχων του δηλαδή και στην εφαρμογή της αποστολής του για την ευρωπαϊκή μέθοδο συντονισμού στην πολιτική ΒΕΤ, δηλαδή επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και βεβαίω με τη συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών. Δεν επικαλύπτει το έργο του με άλλους οργανισμούς ή ευρωπαϊκούς ή εθνικούς ή και Το έργο του ΣΕΝΤΕΦΟΠ υπήρξε και πολύ υψηλής ποιότητας και πολύ αποδοτικό. Θέλω λοιπόν να διατηρήσω αυτά τα υψηλά στάνταρτ, όμως επίσης θέλω να διασφαλίσω ότι ο ΣΕΝΤΕΦΟΠ θα συνεχίσει να παρέχει απαντήσεις στους ε, ηθήνοντες που ασχολούνται με θέματα απασχόλησης, με αυτούς που εγκαταλείπουν ε, πρόωρα την εκπαίδευση, που δεν διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες, αλλά και με αυτούς που διαθέτουν δεξιότητες που όμως δεν έχουν αναγνωριστεί, καθώς και τις επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να ενισχύσουν το e-based learning. Και επίσης θέλουμε να λειτουργήσουμε και ως βάση πρόγνωσης, έτσι ώστε να πετρέψουμε στους ηθήνοντες να ε, σχεδιάζουν και να προσχεδιάζουν το μέλλον. Το Εμείς έχουμε εμπειρία από πρώτο χέρι. Πρωτίστως στην έρευνα των ανθρώπινων πόρων για θέματα επαγγελματικής καταρτήσεως παρακαλούμε, ε, παρακολουθούμε μάλλον το ανακοινωθέν που θα εκδοθεί αργότερα σήμερα παρακολουθούμε την εφαρμογή του, πλαισίου, ε, του ευρωπαϊκού πλαισίου για την εκπαίδευση. Επίσης το Europass το οποίο ήταν 8,7 ε, εκατομμύρια φέτος. Έχουμε και την αξιολόγηση των διαφόρων μορφών ηλεκτρονικής μάθησης. Έχουμε και την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ΕΣΚΟ και για, την εθνική επαγγελματική εκπαίδευση και ούτω καθεξής. Και έχουμε και τη μεθοδολογία ανάπτυξης στατιστικών δικτών για στόχους πολιτικής, για την επαγγελματική εκπαίδευση, για την διαβίου κατάρτιση, βεβαίως σε συνεργασία με τον ΟΣΑ αλλά και με την Ευρωστάτ για να συλλέξουμε ευρωπαϊκά και διεθνή δεδομένα για την VET καθώς και από τις επιθεωρήσεις του ΟΣΑ για τις δεξιότητες των ενηλίκων. Για να συμπεριλάβουμε τα δεδομένα όλα αυτά του ευρωπαϊκού πανοράματος για το 2014 θα προσθέσει και άλλη προσθέμενη αξία στο έργο του οργανισμού. Όπως εξηγούμε και στα σημείωματά μας, είναι να κάνουμε τη γέφυρα μεταξύ των αναγκών της αγοράς και της εκπαίδευσης. Τα βλέπετε όλα αυτά στις ενημερωτικά μας σημειώματα, τα οποία έχετε λάβει όλοι. Και εκεί τονίζουμε την ανάγκη γεφύρωσης μεταξύ της εκπαίδευσης και της απασχολησιμότητας. Και σε αυτά θα ασχοληθούμε και τα επόμενα χρόνια, διότι η αγορά εργασίας απαιτεί οι άνθρωποι να μαθαίνουν διαρκώς την τελευταία δεκαετία έχουν ξεκινήσει πολλά ευρωπαϊκά εργαλεία εντό για να προωθήσουν την λύση αυτή. Η απασχολησιμότητα είναι σημαντική, είναι κρίσιμη για το μέλλον της Ένωσης και η ορατότητα και η σημασία της είναι απαραίτητα για να διασφαλίσουν ότι θα αντιμετωπιστεί η οικονομική κρίση από ένα υπεύθυνο και εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό. Τρεις πτυχές τώρα της κοινή προκλήσεως που θα διέπουν το έργο μας το 2014. Πρώτο, η επαγγελματική εκπαίδευση κατάρτιση των ενηλίκων που ενισχύει ως ΕΝΤΕΦΟΠ έτσι ώστε όλο και περισσότεροι άνθρωποι να έρθουν πιο κοντά στην εμπειρία της εργασίας. Δεύτερο, είναι μια διαρθωμένη προσέγγιση με υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή Συμμαχία Εκπαιδεύσεων και τέλος για το 2014 και πέραν η τεχνική υποστήριξη προς τις χώρες μέλη σε όλες τις πτυχές των ευρωπαϊκών εργαλείων και συνεργειών μεταξύ των εργαλείων. Ο ΣΕΝΤΕΦΟΠ λοιπόν είναι ένας οργανισμός ο οποίος αντιμετωπίζει όλο και αυξανόμενες ανάγκες για την τεχνογνωσία του, ο προϋπολογισμός του αντιμετωπίζει περικοπές. Δεν θα πρέπει όμως να θέσει κίνδυνο την δυνατότητα άσκηση του ρόλου του. Για να επιτρέψει τις χώρες μέλη να συνδράμουν μία γενεά η οποία περνά από κρίση. Εμείς έχουμε το ρόλο να παίξουμε τους διαμεσολαβητές μεταξύ της εκπαίδευσης και της εργασίας, αλλά και της ευρωπαϊκής στρατηγικής και των πραγματικοτήτων των χωρών μελών. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η Πρόεδρο σας ευχαριστώ και δίνω το λόγο τώρα στον Γιώχαν Μενέντες Βάλτες που είναι διευθυντής για την βελτίωση των συνθήκων ζωής και εργασίας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και θερμές ευχές για καλή χρονιά και καλή επιτυχία στις εκλογές. Το 2013 ξεκινήσαμε στο Ίδρυμά μας το νέο τετραετές πρόγραμμα με τίτλο «Από την κρίση στην ανάκαμψη». Βέβαια, ακόμη στην κρίση βρισκόμαστε, αλλά ευελπιστούμε ότι θα μεταβούμε στην ανάκαμψη. Θέλουμε να παρέχουμε πληροφορίες για να, γίνουν, λαμβάνονται αποφάσεις πιο εμπεριστατωμένα για τις πολιτικές. Αυτό είναι ο σκόπος μας. Το 2013 κάναμε το πρώτο βήμα. Εξετάζοντας την κρίση, εξετάσαμε τον αντίκτυπο της κρίσης στη ζωή και την εργασία των εργαζομένων. Κυρίως με τις πανευρωπαϊκές ε, έρευνες που κάναμε σε 14 ευρωπαϊκές χώρες και θα συνεχίσουμε και το χρόνο. Θα πρέπει τώρα να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε την κρίση και τι πολιτικές υιοθετήθηκαν. Εξετάζοντας την κρίση, διαπιστώνουμε από τη δημοσκόπησή μας ότι μειώθηκε η αισιοδοξία των Ευρωπαίων και κάθηκε η εμπιστοσύνη τους προς ε, τους κρατικούς και ευρωπαϊκούς θεσμούς. Μειώθηκε λοιπόν η εμπιστοσύνη στις περισσότερες χώρες μέλη και ιδιαίτερα σε ορισμένες από αυτές ε, καταρακώθηκε. Ένα από τα στοιχεία της έρευνας που δημοσιεύθηκαν και που θα συνεχίσουμε το 2014 αποδεικνύει ότι υπάρχει σύνδεσμος, στενός δεσμός μεταξύ της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς με την παροχή των υπηρεσιών και την ποιότητα των υπηρεσιών που λαμβάνουν από τους κρατικούς θεσμούς. Είναι σημαντικό λοιπόν για τους πολίτες οι, ποιο, οι υπηρεσίες να είναι ποιοτικέ και προσιτές. Έτσι αυξάνεται η εμπιστοσύνη του προ τους, ε, προς τα θεσμικά όργανα. Ξεκινήσαμε την έρευνα μας πέρυσι, θα τη συνεχίσουμε φέτος και επικεντρωνόμαστε σε επιλεγμένες κοινοφελείς υπηρεσίες όπου έχει γίνει περικοπή κονδυλίων, υπάρχουν αυξανόμενες ανάγκες και σε ορισμένες χώρες έγινε μια προσπάθεια για τη βελτίωση της ποιότητας και της πρόσβασης στις υπηρεσίες. Πρόσβαση στη φροντίδα παιδιών, περίθαλψη παιδιών και συνδρομή σε οικογένειες που ζουν υπό επισφαλείς συνθήκες. Κατά το πρώτο της κρίσης, ο δημόσιος τομέας έδειξε μια θεκτικότητα σε ό,τι αφορά την απώλεια θέσεων εργασίας. Αλλά η εξυγίαση δημοσιονομική και η αναδιάρθρωση επηρέασε και το δημόσιο τομέα. Μάλιστα θα δημοσιεύσουμε σχετική έκθεση το 2004 για την αναδιάρθρωση του δημόσιου τομέα και πώς εφαρμόστηκε. Έχουμε διαπιστώσει ότι ένας από τους λόγους της ε, καταστροφής των ε, θέσεων απασχόλησης ε, ήταν η κρίση, η χρεοκοπία που ακολούθησαν, η αναδιάρθρωση, ενώ ταυτόχρονα διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχει πια διαφορά μεταξύ των παλιών και των νέων χωρών μελών. Ενώ, ε, και το offshoring, ενώ κατά την εποχή της διεύρυνσης ήταν εξαπλάσια η διαφορά. Βέβαια η ενεργεία έπληξε περισσότερο τους νέους που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες, αλλά και ο κοινωνικός και κοινωνικός αντίκτυπος της έλλειψης συμμετοχής των γυναικών θα ληφθεί υπόψη στις ερευνές μας. νέοι θα πρέπει να βοηθούν περισσότερο. Θα πρέπει να διευκολυθεί η πρόσβασή τους σε πιο μόνιμες θέσεις απασχόλησης. Γιατί μέχρι στιγμής ε, η ανεργία γιγαντώνεται. Και το θέμα της πρόσβασης στην εκπαίδευση επίσης είναι σημαντικό. Τώρα, πόσες θέσεις απασχόλησης δημιουργήθηκαν για να αντιμετωπιστεί κρίση. Κυρίως ε, εξετάσαμε το θέμα των νέων, ε, της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την πρόσβαση των νέων σε μαθητείες και κατάρτιση. Διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια απόλωση σε ό,τι αφορά τις ε, θέσεις εργασίας και σε ό,τι αφορά τους μισθούς. Οι απώλειες θέσεων είναι κυρίως στη μεταποίηση και στην αυτορικοδομικό κλάδο στις ε, θέσεις ε, χαμηλών και μεσαίων αποδοχών κυρίως. Αυτή η απώλεια δεν αντισταθμίστηκε από βελτίωση στην εκπαίδευση ή αναβάθμιση της ποιότητας των θέσεων απασχόλησης. Υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ των διαθέσιμων θέσεων εργασίας και των, του, μεγάλου κύματος των ανέργων. 40% των επιχειρήσεων δήλωσαν ε, αδυναμία να προσλάβουν τους ε, εργαζόμενους που έψαχναν με ψηλές ειδικότητε, παρόλο που η ενεργεία είναι σε υψηλά επίπεδα. Είχαμε και ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάκαμψη της βιομηχανίας και έχουμε και ένα σχέδιο για τη μεταπητική βιομηχανία στην Ευρώπη και το δυναμικό θέσεων απασχόληση που έχει. Μάλιστα έχουμε και ένα πιλωτικό πρόγραμμα σχετικά θα υποβάλουμε μια έκθεση για τη σχέση μισθού και εργασίας και το σύστημα συλλογικών, επενδύσεων, ε, συλλογικών διαπραγματεύσεων. Συγγνώμη. Ε, θα δημοσιευθεί η έκθεσή μας σχετικά σύντομα μετά την διάσκεψη και του Βίλνιους. Αύξηση της απασχόλησης, βελτίωση των βιωτικών συνθήκων, είναι σημαντικά ζητούμενα του Ιδρύματός μας. Θα συνεχίσουμε τις έρευνές μας λοιπόν και προς αυτήν την κατεύθυνση. Ε, συνεργαζόμαστε και με την όσα. Έχουμε κοινή έρευνα, κοινή έκθεση για τους κοινωνικούς κινδύνους για παράδειγμα. Τώρα για τις περσινές μας επιδόσεις έχουμε ένα προϋπολογισμό γύρω στα 20 εκατομμύρια, όπως θα ξέρετε, 112 ανθρώπους προσωπικό, εφαρμόσαμε τον ε, εκτελέσαμε το 99% του προϋπολογισμού, δημοσιεύσαμε 172 δημοσιεύματα σε μορφή PDF και το πιο σημαντικό είναι ότι στη διαδικασία χάραξη πολιτικών ε, εκδώσαμε 220 έγγραφα πολιτικής, αναλύσαμε ε, 220 έγγραφα πολιτικής στα 50 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης το 2015 θα ενταχθούμε στο δίκτυο ευρωπαϊκών οργανισμών, όπως και η ΩΣΑ. και θέλουμε να βελτιωθεί η διακυβέρνηση των διαφόρων οργανισμών με διοργανική συζήτηση και να εξασφαλίσουμε στενότερη συνεργασία μεταξύ των κοινωτικών οργανισμών και των ειδικών επιτροπών όπως είναι η δική σας. Έτσι θα αναπτύξουμε και καλύτερα συστήματα για να στηρίξουμε και για να ενημερώσουμε καλύτερα και την Επιτροπή Προϋπολογισμών. Σας ευχαριστώ. Η τελευταία μας καλεσμένη, η κυρία Μαγκλέν Σερμπάν, η Διευθύντρια του Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Πρόεδρε, εγώ θα ήθελα, όπως και οι συνάδελφοί μου, να σας ευχηθώ σε εσά αλλά και σε όλους τους ευρωβουλευτές ε, υγεία και επιτυχία. Ε, ελπίζουμε πως μετά το καλοκαίρι θα υπάρξει και η ε, πολυπόθητη ανάκαμψη. Ως EDF θα σας μιλήσω για τον προπολογισμό μας που προέρχεται από το κονδύλιο που αποκαλείται Global Europe. Ε, επιτυχείς πολιτικές ε, λοιπόν και διάδοση αυτών και αυτός, μπορούμε σήμερα λοιπόν να σας πούμε ποια είναι τα επιτεύγματά μας προς αυτή την κατεύθυνση. Σε σχέση με το 2013 και προσλάβοντας για το 2014 καταρχήν Βρίσκομαι σε μια, στη θέση να αναφέρω πως το 2013 είναι το τελευταίο ε, έτος των ε, μέσων προοπτικών για τη τετραετία 2010-2014. Έχουν υπάρξει κάποια επιτεύγματα, ενώ το 2014 είναι νέα τετραετία 14 με 17 και έχει προγραμματιστεί σύμφωνα με τη στρατηγική TF 2020 που υιοθετήθηκε τον περασμένο Νοέμβριο από το Διοικητικό Συμβούλιο. Γιατί το Global Europe είναι σημαντικό και πιστεύουμε πως έχει νόημα να είμαστε ακόμα πιο δραστήριοι ε, γιατί ακριβώς η αλληλεξάρτηση των χωρών σε όλο και περισσότερου τομεί πολιτική ήδη απαιτεί άνευ προηγουμένου συνεργασία οι σχέσεις ανάμεσα στις κυβερνήσεις και την Ένωση αλλά και την Ένωση με χώρες που δεν είναι μέλη της Ένωσης, αλλά και είναι εξίσου σημαντική η συνεργασία με τα χώρες εκτός Ένωσης. Η διαχείριση πληροφοριών ανάμεσα ε, για τις διάφορες πολιτικές, εθνικές ε, χώρες ή διεθνείς είναι πιο περίπλοκη και είναι πολύ σημαντική όμως για τη βιωσιμότητα και την ε, σταθερότητα και γι' αυτό και πιστεύω πως το παγκόσμιο ενδιαφέρον δεν, δεν συμφέρον μάλλον δεν θα πρέπει να είναι μάλλον το γενικό συμφέρον δεν θα πρέπει να είναι δευτερεύον σε σχέση με τις προτεραιότητές μας. Ε, χθες κοιτούσα τα Euronews και τι είδα, αναταραχές στην Ουκρανία, ειρηνευτικές ε, διαπραγματεύσεις για τη Συρία, ε, εντάσεις στο Λίβανο και στην Αίγυπτο, προσχώρηση της Τουρκίας ε, και της Σερβίας στην Ένωση. Ένταξη. Αυτά. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Πώς λοιπόν μπορεί κανείς να δουλέψει όταν Ε, τόσο, σε, σε χώρες όπου επικρατεί τόσο μεγάλη αστάθεια. Αυτή, αυτό είναι το βασικό μας ε, ερώτημα και πιστεύουμε πως η δουλειά μας για την ανάπτυξη εργατικού δυναμικού είναι βασική για την ανάκαμψη αυτών των χωρών. Και αν στην Ευρώπη θεωρούμε δεδομένη τη δημοκρατία και τις αξίες αυτής, στις χώρες αυτές έχουν νόημα οι αξίες οι δημοκρατικές και έχει νόημα το να συνεχίσουμε να τις βοηθούμε. Γι' αυτό και πιστεύουμε εντόνως ότι η ιδιοποίηση και η συμμετοχή αυτών των χωρών, ε, των πολιτικών και ε, είναι προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη, συμβάλλει στην αύξηση της ανθεκτικότητας των εθνικών συστημάτων τους, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, αλλά και σχηματίζουν τις δυνατότητες όλων αυτών των εθνών και των οργανισμών τους να αντιμετωπίσουν προκλήσεις αλλά και την αστάθεια και την αβεβαιότητα. Γι' αυτό και προσέχουμε πάρα πολύ ε, όσον αφορά την εκμάθηση πολιτικής. Γιατί θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι εκεί όπου επικρατεί μεγάλη αστάθεια είναι σημαντικό να διευρυνθεί η συμμετοχή των φορέων και γι' αυτό και η εργασία του ETF στην πολυεπίπεδη διακυβέρνηση είναι πολύ σημαντική και θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για την προσωπική σας υποστήριξη και για την στήριξη γενικότερα της Επιτροπής Απασχόλησης για τις δραστηριότητε πολιτικής που ασκούμε τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα για τις χώρες της Μεσογείου, τις αραβικές χώρες όπου ξεκινήσαμε στο Αμάν το 2012 μετά στην Μασαλία το 2014 και το ίδιο κάναμε και για τα Δυτικά Βαλκάνια τον Οκτώβριο του 2012. Είναι πολύ σημαντικό αυτό ώστε οι ηγέτες πολιτικοί και το κοινοβούλιο να εμπλέκονται σε όλες αυτές τις συζητήσεις και είναι πολύ σημαντικό για τη δημιουργία θεσμών έτσι ώστε να είμαστε βέβαιοι πως και οι πολιτικές αυτές θα εφαρμοστούν κιόλα, δεν θα υιοθετηθούν απλά στις διάφορες περιφέρειες. Επίσης εργαζόμαστε για τη διακυβέρνηση σε υπό σε, περιφερειακό επίπεδο σε διάφορες χώρες και θα το είδατε και στα έγγραφα που σας ενεμήθηκαν, ακόμα και σε επίπεδο δηλαδή σχολείων δουλεύουμε, έτσι ώστε να είμαστε βέβαιοι πως όλοι θα είναι σε θέση να ε, εφαρμόσουν τις πολιτικές, ε, αναζητούμε τις καλές πρακτικές ώστε να σχηματίσουμε ε, τέτοιες πολιτικές όταν αυτό χρειάζεται. Πιστεύουμε εντόνως δε ότι η εργασία μας για την σε δεξιότητες, για την απασχόληση και την δυνατότητα απασχόλησης θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν καλύτερες ευκαιρίες για τους πολίτες των χωρών αυτών, έτσι ώστε να αναζητήσουν το μέλλον τους στις χώρες τους. Αυτό είναι η πρώτη μας και η σημαντικότερη μας εντολή και καθήκον, αλλά ε, ξέρουμε ότι υπάρχει και κυκλική μετανάστευση, έτσι ώστε αν υπάρχει κινητικότητα βορράς, νότο, νότος, βορράς, εν πάση περιπτώσει γεωγραφικά, το γεωγραφικό σκέλος δεν έχει τόση σημασία, πάντως να μπορούμε να εξασφαλίσουμε για τους πολίτες του μέλλοντος, το μέλλον τους στη χώρα τους ή όπου και αν πάνε, γιατί ε, ξέρετε και ότι η μετανάστευση πολύ, ε, πολύ συζητείται το τελευταίο καιρό στην Ευρώπη. Το κάνουμε αυτό ε, από το 2013 και για τις χώρες όπου υπάρχει ε, μια βόμβα δημογραφική. 60 εκατομμύρια θέσεις απασχόληση θα χρειαστούν τα επόμενη αιτία εκεί. θα πρέπει λοιπόν να βρούμε Ε, θέλουμε λοιπόν να προετοιμαστούμε. Ε, μιλάμε λοιπόν για το 2014. Δεν είναι σημαντικό, είναι σημαντικό να θυμηθούμε ναι, ότι θα γιορτάσουμε τα 20 μας χρόνια. Αλλά όταν ο πρόεδρος της Επιτροπής αποφάσισε να φτιάξει το ETF, ο Ζακ Τέλορ μαζί με τον επικεφαλής του επιτελείου του, τον Πασκάλ Λαμή, και έβαλε στο τραπέζι όλες τις προτάσεις, έλαβαν υπόψη το γεγονός ότι αν πέσει το τείχος του Βερολίνου θα χρειαστούν λύσεις για αυτές τις χώρες. Και γι' αυτό και όταν μιλάμε για τα νεα κρατημέλη είμαστε ευτυχείς και περήφανοι που συμβάλαμε κι εμείς. Αλλά το 2014 είναι και η εκατονταετία από τον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο που ξεκίνησε στο Χισεράγευο. Ακόμα ένα μέρος του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Κατάρτισης και ελπίζουμε πως όλες αυτές οι υπερχόμενες επέτειοι του παγκοσμίου και του οικονομικού χάους που υποκράτησε μετά από το πρώτο παγκόσμιο θα, χρησιμοποιήσουν, θα χρησιμεύσουν ως υπενθυμίσεις για τους ηγέτες αλλά και για τους πολίτες ότι τα προβλήματα θα πρέπει να τα διαχειριστούμε. Θα πρέπει να τα διαχειριστούμε και μετά το 2014 και αργότερα ε, την παγκοσμιοποίηση έτσι ώστε να είναι αποδοτική για τους περισσότερους και όχι μόνο για ορισμένους. Και χθες το βράδυ Ακούσαμε με μεγάλη χαρά και περιφάνεια για το ETF. Έμαθα λοιπόν ότι δύο Υπουργοί Εξωτερικών, και δεν είναι νομίζω τυχαίο, προέρχονται από τις ίδιες χώρες, Γαλλία και Γερμανία, ο κύριος Λοράν Φαμπιούς και ο κύριος Μάιερ αποφάσισαν να κατέβουν στις ευρωεκλογέ στη δημοκρατία της Μολδαβίας και της Γεωργίας, δύο χώρες του ETF. για να συζητήσουν με τους πολίτες των χωρών αυτών για τις αξίες της Ευρώπης. Γι' αυτό πιστεύουμε πως η Ευρώπη, ε, Global Europe έχει νόημα και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να την προωθήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία μου. Ευχαριστώ τους τέσσερις διευθυντάς. Δεν είμαστε πια πολύ άριθμοι, βλέπω όμως ότι όλοι επιθυμούν να λάβουν τον λόγο η Σάρα Πάρκιν που είναι η εμπειρογνώμων στο Συμβούλιο του ETF επιθυμεί επίσης να λάβει το λόγο αλλά σας παρακαλώ πραγματικά συντομότατα έστω να προλάβουν και οι βουλευτέ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ έχω συντάξει ένα έγγραφο που νομίζω ότι έχουμε, έχει διανεμηθεί σε όλα τα μέλη της Επιτροπής και δίνει μια σύντομη περίληψη του πώς διαρθρώνει τις αποφάσεις του το ETF. Περισσότερο αυτό και λιγότερο το τι ακριβώς κάνει. Το πρόγραμμα εργασιών για το 2014 επίσης διαλαμβάνεται εκεί. Το πιο σημαντικό γι' αυτό είναι ότι περάσαμε δύο γύρους τη διαδικασία του Τουρίνου, δηλαδή οι χώρες μέλη εξετάζουν τα στοιχεία που βρίσκονται και αυτό καθιστά ευκολότερο το έργο του ETF να καταστρώσει δηλαδή τις προτεραιότητές του κομμένες και ραμμένες όπου είναι απαραίτητος όπως εξήγησε η κυρία Σερμπάν. Πορτρέζω λοιπόν της κάθε χώρας που τους επιτρέπει μετά να ανακτήσουν την κυριότητα των πολιτικών και δομών που θεσπίζουν και επίσης επιτρέπει την κοινή χρήση των καλών πρακτικών που επίσης είναι σημαντικό. Το ETF επιθυμεί να συμμετάσχουν περισσότερες χώρες στην διαδικασία του Τουρίνου και επίσης και η ποιότητα να αυξηθεί με οδηγούς και άλλα εργαλεία που όπως εξήγησε η κυρία Σερμπάν γιατί η διαχείριση, η διακυβέρνηση είναι πολύ σημαντική σε όλα τα επίπεδα και είναι πολύ σημαντική επίσης για την τοπική ανθεκτικότητα, την ανθεκτικότητα δηλαδή των τοπικών κοινωνιών. Οι προϋπολογισμοί που διατίθενται σύμφωνα με τους στόχους, τους τρόπους παρεμβάσεων και, τους, λειτουργίε. τις υπήρξε σημαντική βελτίωση στην σύγκριση εφαρμογής των στρατηγικών προγραμμάτων και δημιουργίας των προϋπολογισμών. Και έκαναν πλήρη έλεγχο πέρσι οι λογιστές εγώ ε, για μένα προσωπικά πηγαίνω στη συνεδριάσεις του ε, Συμβουλίου. Έχω συμμετάσχει στην εκπόνηση της Μεσοπρόθεσμης Στρατηγικής και του Προγράμματος Εργασιών 2014. Ε, απίθυνα το λόγο σε μία από τις διασκέψεις για την βιωσιμότητα και καινοτομία και νομίζω ότι πολύ περισσότερα πράγματα μπορούν να γίνουν για να μεταρρυθμιστούν κάποιες από τις ε, άκαμπτες κάπως συνήθειες του συστήματος VET, VET των επαγγελματικών καταρτήσεων δηλαδή. Και όπως το παρελθόν, βασικός μου στόχος, γιατί εγώ είμαι ε, μέλος του Συμβουλίου που δεν ψηφίζει, ο βασικός μου στόχος λοιπόν είναι για οργανωτικά θέματα και βεβαίως βασίζομαι στην ε, σχετική εμπειρία που έχω. Για το μέλλον νομίζω ότι το Κοινοβούλιο αλλά και για άλλες διευθύνσει θα πρέπει να σκεφτούν σοβαρά την ανάγκη διασφάλισης της senior expertise στο ETF σε δύσκολες περιόδους για την απασχόληση. Γιατί υπάρχει κίνδυνος να χαθεί η τεχνογνωσία αυτή. Το Νοέμβριο σημειώνουμε, εορτάζουμε την 20 αιτία και είναι σημαντικό να διατηρηθεί και να προωθηθεί το έργο του ETF, όχι μόνο μέσα στην Ένωση αλλά και στις ε, χώρες εταίρους. Τελευταίο, τελευταίο κυρία Πρόεδρε, γιατί είναι για το μέλλον και είναι και πολιτικό θέμα. Η καιρή θα είναι δύσκολη στο μέλλον. Το ETF και η δουλειά που κάνει και βεβαίως και το έργο και ορισμένων άλλων οργανισμών είναι να προσφέρουν ένα σημαντικό ουδέτερο έδαφος. Σας ευχαριστώ πολύ. Διακόπτη η Ευγενώση Πρόεδρος, τον κύριο το λόγο κύριο Σέρκας. Γιατί όλοι θέλουν το λόγο. Κύριο Σέρκας. Τηλεγραφικά κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διευθυντές των Ινστιτούτων και Ιδρυμάτων και Οργανισμών και να τους πω ότι μπορεί να μην είμαστε πολλοί ευρωβουλευτές παρόντες στην αίθουσα, αλλά σας διαβεβαιώ ότι εκτιμούμε ιδιαίτερως ε, τις προσπάθειες και το έργο σας. Και απόδειξη αυτές οι προσκλήσεις ε, για συμμετοχή. Θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση κοινή προς όλους. Πώς καταφέρετε με αυτή το πάγωμα του προϋπολογισμού θα καταφέρετε να συνεχίσετε τις ε, εργασίες σας ενώ όλο και περισσότερο έχουμε ανάγκη από τις μελέτες σας, τις έρευνές σας και την αξιοποίηση, αξιοποίηση των βέλτιστων πρακτικών. Και από τον οργανισμό του Bilbao θα ήθελα να μάθω τι γίνεται με τη στρατηγική για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία. Από το ΣΕΝΤΕΦΟΠ θα θέλαμε να μας πείτε τι γίνεται με τη διτή επαγγελματική κατάρτιση. Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Για το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωση και εργασία, Πολύ σωστή εκτίμηση ότι παρόλο που είμαστε εν μέσω τη κρίση, φοβόμαστε ότι ο στόχος ε, κατά εξάλληψη της φτώχειας θα επισκιαστεί στη Γενική Στρατηγική του 2020. Επίσης έχουμε πρόβλημα με την ενεργεία των νέων και με τη στεγαστική πολιτική στην Ευρώπη. Αυτά ευχαριστώ. Σημαντικό είναι και το έργο του Ιδρύματος Επαγγελματικής εκπαίδευση, ε, Όπως σωστά είπατε, δεν είμαστε απομονωμένοι νησί ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε πολλές χώρες ε, με τις οποίες συνεργαζόμαστε, με τις οποίες έχουμε διάλογο και πολλές υποχρεώσεις απέναντι τους. Ε, κύριε Χιούς, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους τέσσερις διευθυντές και την εμπειρογνώμονα για τις ομιλίες τους και να επαναλάβω αυτό που είπε ο Αλεχάνδρο, μην εκλάβετε την απουσία των βουλευτών από τη συνεδρίαση ως έδειξη αδιαφορίας ε, ή απαξίωσης ε, των οργανισμών σας. Εκτιμούμε ιδιαίτερα στο έργο των οργανισμών και ιδρύματων σας. Και αναφέρθηκε από το Διευθυντή του Δουβλίνου ότι πολλά έγγραφα και δικά μας και δικά σας ε, αναφέρουν το έργο του Eurofound. Επίσης και για την όσα για τον Οργανισμό Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία. αν είχαμε εγκαίρως μια πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως είπατε, για νέα στρατηγική για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία, θα ήταν πολύ χρήσιμο. Αλλά μετά από τόσα χρόνια χρησιμοποιούμε δικαιολογίες και προσχήματα για να αποφύγουμε την εφαρμογή της νέας στρατηγικής. Επίσης, ποια είναι η γνώμη της Διευθυντηρίας του οργανισμού του Μπιλμπάου για αυτή την κολυσιεργία. Εγώ ασχολούμαι ιδιαίτερα με τους οργανισμούς του Μπιλμπάου και του Δουβλίνου γιατί λαμβάνω υπόψη τις θέσεις τους στις εκθέσεις που υποβάλλω στην Επιτροπή. Έχω μερικές παρατηρήσεις λοιπόν και κάποιες ερωτήσεις. Για τον Μπιλμπάου. Χαιρετίζω το έργο σας σε περιοχές που υπάρχει κίνδυνος ε, ή μάλλον πιθανότητα εμφάνισης κινδύνου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να ληφθεί υπόψη και στο νομοθετικό έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και στο παρελθόν ο ρόλος του Μπιλμπάου ήταν πολύ χρήσιμο στον εντοπισμό ε, αναφιόμενων κινδύνων. Επίσης, ε, για, τις, ε, για τους επανειλημμένους τραυματισμούς στην εργασία, το έργο του ΩΣΑ, μειοσκελετικές παθήσεις, πολύτιμη συμβολή τους στα θέματα αυτά. Επίσης, ψυχοκοινωνική κίνδυνη. Χαίρομαι που αναφέρθηκε η λήψη υπόψη και του θέματος αυτού του ψυχοκοινωνικών κινδύνων στο σχέδιο εργασίας 15-16. Αν δεν κάνω λάθος και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει Είχε υποσχεθεί πριν από 20 χρόνια να υποβάλει μια πρόταση για τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους, δυστυχώς ακόμη την περιμένουμε σε ό,τι αφορά τον οργανισμό του Μπιλμπάου. Κάνετε κάτι και μέσω του δικτύου σας για να καταμετρήσετε το κίνδυνο, ε, την επίδραση μάλλον των μέτρων λιτότητας ε, στην ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων στην Ευρώπη. Ίσως είναι κάπως πρόωρο αυτό. Ρωτιέμαι όμως είναι στα σχέδιά σας για το μέλλον. Για τον οργανισμό του Δουβλίνου. Μετά από πολλές πιέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρχές Οκτωβρίου ανήγγειλε το νέο πίνακα επιδόσεων, το νέο βαθμολόγιο το κοινωνικό στα πλαίσια της ΟΝΕ. Το Ίδρυμα του Δουβλίνου θα διαδραματίσει κάποιο ρόλο τροφοδοτώντας με πληροφορίες την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υποβολή του νέου πίνακα επιδόσεων. Ευχαριστώ. Παρότι αργά θέλω να θέσω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη αφορά την οργανισμό όσα ε, ε, για τη στρατηγική της ασφάλειας και της υγείας στο χώρο εργασίας. ποια, είναι η φύση του διαλόγου σήμερα συγκεκριμένα ανάμεσα στον οργανισμό και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενώ προφανώς υπάρχει πολιτικό μπλοκάρισμα ε, για να ξεκινήσει αυτή τη στρατηγική και να την προωθήσει Κομισιόν και έχετε γνωρίζετε μάλλον ποια είναι η συμβολή που μπορείτε να κάνετε στην κατάλληλη στιγμή. Ευχαριστώ που αναφέρατε και το θέμα του στρες, που είναι ένα θέμα το οποίο έχει πολύ απασχολεί στην Επιτροπή μας όταν ζητήσαμε την αναθεώρηση και την έναρξη αυτής της στρατηγικής. Το Σεντιφόπ νομίζω πως εκδώσατε μια πολύ σημαντική μελέτη όσον αφορά τις προδιακυβεύματα για τους ε, κατώτατους μισθούς μετά από τις σχετικές πολιτικές συζητήσεις. Ε, α, σας ευχαριστώ κυρία Πάτριν που συμμετείχατε σε αυτήν την ακρόαση, αλλά εν πάση περιπτώσει το σημειώνω ότι δεν κάθεστε μέχρι το τέλος. Ε, εντάξει. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, έγινε αυτή η συζήτηση για το ε, τους μισθούς μετά από τη συμφωνία του συνασπισμού στη Γερμανία. Εσείς, εσείς συνδεθήκατε με αυτή τη συζήτηση και ναι, με ποια μορφή για τους επόμενους, τις επόμενες φάσεις προβληματισμού της Κομισιόν. Λοιπόν, θα είμαι πολύ αυστηρή στρατιωτική. Θα έχετε δύο λεπτό καθένας για να απαντήσετε στα ερωτήματά μας. Ξέρω ότι μπορείτε να είστε πολύ αποτελεσματικοί. Και θα ξεκινήσουμε με την ίδια σειρά, δηλαδή με την Κρίστα Σεδλατσέκ. Σας ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ ακόμη μια φορά για τη στήριξη που μας δίνει η Επιτροπή σας και βεβαίως μπορώ να σας δώσω ποια ήταν η ανταπόκριση. Εμείς ε, υποφέρουμε από τις περικοπές, αλλά πιστεύω πως όλοι οι διευθυντές που είμαστε εδώ σήμερα ξέρουμε πως είναι καθήκον μας να οργανώσουμε τη δουλειά μας με τρόπο ώστε να μπορέσουμε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μόνο όμως για να σας δώσω ένα παράδειγμα, το δίκτυο του οργανισμού που βασίζεται στα 28 κρατημέλη αυτή τη στιγμή ε, πάσχει γιατί κάποια μέλη του δικτύου δεν είναι σε θέση να πάνε σε αποστολές να παρακολουθήσουν τις συνεδριάσεις μας. Και δεν είναι η Γερμανία ούτε η Σουηδία. Είναι οι χώρες όπου πραγματικά θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε και να στηρίξουμε στο στρατηγικό προγραμματισμό. Αυτό βεβαίως το αισθανόμαστε. Και πρέπει να πω ότι βεβαίως περιλαμβάνεται και το θέμα της κρίσης, το αντίκτυπο της κρίσης στην ασφάλεια και την υγεία σε όλα τα επίπεδα, αλλά και σε σχέση με τις δημογραφικές αλλαγές, γιατί βλέπουμε ταυτόχρονα πως τώρα και στο μέλλον θα είναι πάρα πολύ κρίσιμη σημασία για την ευρωπαϊκή οικονομία να διατηρηθεί σε υγιή κατάσταση το εργατικό δυναμικό και σε ασφαλή κατάσταση. Μιλάμε για την παράταση της εργασιακής ζωής και εδώ μπορεί κανείς να έχει πολύ στρες και αυτή είναι και η βάση της δουλειάς μας για το μέλλον. Δεν είμαστε βέβαια ευτυχεί καθόλου που δεν υπάρχει ευρωπαϊκή στρατηγική για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία. Ωστόσο, έχουμε αρκετά καλή σχέση με την Κομισιόν και βεβαίω δεν είναι μόνο με το τμήμα. Ε, ε, ξέρουμε όμως ότι υπάρχει επιθυμία σε ανώτερα επίπεδα για να υπάρξει μια νέα, εκπονηθεί μια νέα στρατηγική και έξω ότι τον Απρίλιο θα γίνει η ανακοίνωση για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία. Συνεργαζόμαστε λοιπόν και προσπαθούμε να διατηρήσουμε όσο γίνεται τη στήριξη, αλλά φυσικά δεν είναι δική μας αυτή η απόφαση. Τώρα, επανέρχομαι στη Γερμανία και την νομοθεσία της. Ε, Ήμουν στην Γερμανία ε, προ καιρού έχουμε πολύ καλές σχέσεις συνεργασίας, ε, νομοθεσία ε, κατά του στρες ε, συντάσσεται εκεί. Ήταν εντυπωσιακό το γεγονός ότι τουλάχιστον οι πληροφορίες του οργανισμού μας χρησιμοποιούνται για να συζητηθεί το κατά πόσο χρειάζεται τέτοια νομοθεσία στη Γερμανία. Είναι επίμαχο το θέμα και ήμουν εκεί πριν τις εκλογές και ε, έχω στενούς δεσμούς με το Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνης. Ξέρω πως η κατεύθυνση αλλάζει και υποσχέθηκα ότι τον Αύγουστο που θα έχουμε την παγκόσμια διάσκεψη στη, στη Φραγκφούρτη θα έχουμε επιπλέον στοιχεία για τη Γερμανία. Ευχαριστώ πολύ κυρία Διευθύντρια. Εσείς τώρα, δύο λεπτά. Ναι, πολύ σύντομα. Σε ό,τι αφορά τις περικοπές στον προϋπολογισμό, αυτή είναι η πραγματικότητα της σήμερων. Όμως κάνουμε σημαντική προσπάθεια για την ευκαμψία και τον εξορθολογισμό των ανθρώπινων πόρων μας που διδιαθέτουμε διαθέτουμε στα πλαίσια του ΣΕΝΤΕΦΟΠ. Παράδειγμα, παρόλο που υπάρχουν δυο μονάδες, μία για στρατηγικές πολιτικής και άλλοι για την ενισχυμένη συνεργασία, οι εμπειρογνώμονες πηγαίνουν από τη μια μονάδα στην άλλη για να κάνουν έρευνα και προσανατολισμό. Δηλαδή ήδη μοιραζόμαστε τη γνώση ανάμεσα στις δύο μονάδες. Περισσότερο από αυτό όμως εντείνουμε τη συνεργασία μας για παράδειγμα με το ETF. Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα διεξαγάγαμε κοινό σεμινάριο και θέλουμε να συνεχιστεί και να ενταθεί αυτή η συνεργασία. Έτσι λοιπόν μέσα στους περιορισμούς του προϋπολογισμού προτιθέμεθα να κάνουμε πληρέστατη χρήση των διαθεσίμων πόρων εποφελία των Ευρωπαίων πολιτών. Βέβαια πρέπει να δώσουμε αξία σε κάθε είδους εκπαίδευση και την επίσημη και την μη επίσημη εκπαίδευση. Και αυτά είναι σημαντικά, σημαντικές πτυχές και για την επίτευξη των στόχων του ορίζοντα 2020 και θα θέλαμε όλες οι χώρες μέλη να κινηθούν προς την κατεύθυνση αυτή. Βεβαίως δεν κινούνται όλες με την ίδια ταχύτητα στην εφαρμογή των ευρωπαϊκών εργαλείων. Αυτό που θέλουμε εμείς είναι να εντείνουμε την χρήση των πόρων και τη συνεργασία με τις χώρες μέλη, έτσι ώστε να ξεφύγουμε από το μικρο και να πάμε στο μακροοικονομικό επίπεδο. Ευχαριστώ. Εσείς τώρα κύριε Μενέντες Βαγιές, σύντομα, μειώσεις προϋπολογισμού, μειώσεις και προσωπικού βεβαίως και έχουν επιπτώσεις, θα ήταν αφελές να πω ότι δεν έχει, ότι θα ήταν ορθό, μιας και έχουμε φτάσει στις 40 40 ώρες εργασίας ότι θα είναι πιο εύκολα. Έχω, κάνουμε όμως συνέργειες, περισσότερη έρευνα in-house με τον επιχειρησιακό προϋπολογισμό που έχουμε. Έχουμε βέβαια σημαντικές δυνατότητες. Τώρα, θα και με τη φτώχεια, τον κοινωνικό αποκλεισμό, με καλύτερη κατανομή για την στέγη επίσης. Θέλουμε ένα πρόγραμμα για τα επόμενα χρόνια και αρχίζουμε ήδη. Για τα σχόλια τώρα του κυρίου Χιούς για το κοινωνικό βαθμολόγιο. Ένας από τους σημαντικούς δείκτες εκεί είναι οι ανάγκες. Υπάρχουν και οι υποδείκτες που χρησιμοποιούμε για την χρήση από την επιθεώρηση των συνθήκων εργασίας και ούτω καθεξής. Και τέλος η κυρία Μπερές είπε για τους μισθούς Αυτά θα δημοσιευθούν. Έχουμε επαφές και με τα Υπουργεία στο Βίνιους αλλά και με την Κομισιόν. Βεβαίως και η συζήτηση στη Γερμανία παίζει ένα ρόλο. Βέβαια η Γερμανία έχει το μεγαλύτερο ποσοστό ανθρώπων κάτω από τα 60 και να δούμε ποιε θα είναι οι διαφορετικέ πολιτικέ επιλογέ, αν θα συντονιστούν οι πολιτικέ ή όχι κτλ. Εμεί παρουσιάσαμε ορισμένα ενδιαφέροντα αποτελέσματα για την σχέση μεταξύ μισθών, γιατί υπάρχουν και ειδικέ συστάσεις για χώρες και είναι πολύ ενδιαφέροντα τα ευρήματα και ότι υπάρχουν, υπάρχει βεβαίως ε, ε, σχέση μεταξύ των ε, μισθών και των αποτελεσμάτων. Ευχαριστώ, αλλά αυτές οι ανησυχίες εμπίπτουν σε άλλες συζητήσεις για τις αρμοδιότητες του Eurofund και είναι σημαντικό να έχουμε τις πληροφορίες από τη βάση δεδομένων για να, μπορούμε, για να μπορέσουμε να συμβάλλουμε στη συζήτηση. Από εδώ και πέρα θα συνεχίσουμε στα αγγλικά γιατί πρέπει να φύγουν οι διερμηνείς.